con la reunión de la comisión punto número 13 παρουσίαση μιας μελέτης για την αλληλεία ανεπαρκούς τεκμηρίωσης στα ευρωπαϊκά ύδατα όπως ξέρετε ζητήσαμε να γίνει αυτή η μελέτη με στόχο να έχουμε μια τεκμηρωμένη βάση για τους ε, αλληλευτικούς πόρους η υπηρεσία ε, η αρμόδια γι' αυτό ανέθεσε τη μελέτη σε ένα Ινστιτούτο στο νέο Βασίλειο. Σας έχει διανεμηθεί η μελέτη αυτή. Οπότε ε, να καλωσορίσω θερμά στην Επιτροπή μας τους δύο ε, συντάκτες της έκθεσης Ryan και Ken και θα σας δώσω στο λόγο θα σας δώσω το λόγο για να μας παρουσιάσετε το κείμενό σας, την έκθεσή σας, τη μελέτη σας και μετά θα το συζητήσουμε. Ανεφετέρων, σας ευχαριστώ και πάλι, σας καλωσορίζω και ο κύριος Μπράιαν έχει το λόγο. Ο κύριος Ομπράιαν. Ο κύριος Ομπράιαν. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Ομπράιαν. Ευχαριστούμε την Επιτροπή σας για την ευκαιρία να καταρτήσουμε αυτή την έκθεση. Νομίζω επειδή έχει γίνει πολύ ερευνητική εργασία, ήταν κατάλληλη στιγμή. Εξετάζουμε τα ενωσιακά ύδατα για να υπάρξει μία μελέτη σε βάθος για το θέμα αυτό. Βόρειο, Ανατολικός, Ατλαντικός, Βαλτική, Μεσόγειος, Εύξηνος. Η εργασία είχε δύο τμήματα. Πρώτον, να μελετήσουμε τις ε, επιστημονικές συμβουλές που δίδονται για την αλία στην Ένωση και να καθορίσουμε τα αλλιεύματα και τις εκφορτώσεις για να μπορέσουμε να ε, κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις ε, αλλιεύσεις. Επίσης θέλαμε να εξετάσουμε και να μελετήσουμε τις μεθόδους για την ε, δημιουργία και χορήγηση επιστημονικών συμβουλών. Και επίσης να κοιτάξουμε εναλλακτικές ε, μεθόδους που υπάρχουν στην Αμερική, τον Καναδά, την ε, Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και να ασχοληθούμε και με τη, τα στοιχεία από το GFCM Λοιπόν, ε, ποιοι είναι οι τομείς, ε, ποια είναι η αποτίμηση των, ε, της αλληλείας, ποιες είναι οι αλλιεύσεις όπου δεν έχουμε στοιχεία, πώς τις μελετάμε και τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η έκθεση εξετάζει όλα αυτά τα κεφάλαια. Θα δώσω το λόγο στον Will που θα σας μιλήσει για τα κεφάλαια αυτά ένα-ένα και θα απαντήσω ρωτήσω στο τέλος. Παρακαλώ. Ωραία. Δεν θέλω σε αυτή τη φάση να μπω σε πολλές λεπτομέρειες. Να σας κάνω μια γενική παρουσίαση. Ένα πρώτο ερώτημα. Για ποιο στόχο να κάνουμε ε, αποτίμηση ή εκτίμηση των αποθεμάτων. ούτως ώστε να υπάρχει βάση για ε, σκόπιμη διαχείριση. Θέλουμε ενημέρωση για την κατάσταση των ε, αποθεμάτων σε σχέση με τους στόχους διαχείρισης και πληροφόρηση για την επίπτωση των διαφόρων διαχειριστικών επιλογών. Πώς θα επηρεάσουν την μελλοντική κατάσταση των αποθεμάτων. Η πληροφόρηση λοιπόν αυτή σχετίζεται και με τους στόχους της αλληλευτικής διαχείρισης και τα μέσα που θα έχουν στη διάθεσή τους ε, οι διαχειριζόμενοι την αλληλεία. Ε, η διαχείριση της αλληλείας γίνεται με βάση την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Στις περιοχές του βόρειο-ανατολικού βόρειο Ατλαντικού και της Βαλτικής καθορίζονται ποσοστώσεις ή ΤΑΚ, μέγιστη επιτρεπόμενη αλίευση η μέγιστη επιτρεπόμενη απόδοση βασίζεται σε σημεία αναφοράς. Προηγουμένως είχαμε απλώς ορισμένα όρια που απαιτούσαν ε, διαφορετική ε, τεκμηρίωση. Ενώ στη Μεσόγειο, όπου η διαχείριση βασίζεται στον, ε, στη ρύθμιση των προσπαθειών και όχι σε τάκ, θα έπρεπε η προσπάθεια ανααλίευμα να συνδυαστεί με τα στοιχεία αυτά. Λέω πολλά για αυτό το θέμα, τη σχέση μεταξύ των αναγκών της διαχείρισης και τις απαιτήσει της εκτίμησης, γιατί είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι πάει να πει ανεπαρκώς τεκμηριωμένη αλία και να δούμε τι επιλογές έχουμε. Επαναλαμβάνω. Οι ανάγκες της διαχείρισης ε, καθορίζουν τον τόπο των στοιχείων, αλλά και αντίστροφα, όπου είναι περιορισμένα τα στοιχεία, αυτό έχει επιπτώσει στις διαχειριστικές επιλογές. Στη μελέτη μας συζητάμε την αποτίμηση των αποθεμάτων. Θέλουμε λοιπόν να αποτιμήσουμε το μέγεθος των αποθεμάτων. Αλλά στα πλαίσια γενικότερα της διαχείρισης ίσως χρειαζόμαστε και περισσότερες επιπτώσεις για τις επιπτώσεις της αλληλείας στο ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα. Αυτό είναι εκτός ε, στόχου της έκθεσής μας. Εμείς κυρίως ασχολούμαστε με την αποτίμηση των αποθεμάτων. Αν μιλήσουμε για, αυτές τις, για αυτή την αλληλεία, την ε, αλληλεία ανεπαρκούς τεχμηρίωσης, τι είναι η αλληλεία όπου έχουμε επαρκή και μάλιστα πλούσια στοιχεία. Είναι τα ίδια αλληλείας όπου μπορούμε να έχουμε στοιχεία και για το μέγεθος ε, των ε, αποθεμάτων και για την θνησιμότητα ε, των αλλιευμάτων. Δηλαδή έχουμε στοιχεία και για τις εκφορτώσεις και για τις απορρίψεις. Έχουμε επίσης στοιχεία για το ποιοι είναι οι ρυθμοί ορίμανσης, οι ρυθμοί ανάπτυξης και μοντέλα εξέλιξης του πληθυσμού. Έχουμε λοιπόν σε αυτή τη φάση, σε αυτές τις περιπτώσεις, πάρα πολλά στοιχεία για αυτά τα είδη των αλλευμάτων. Μία ε, αλία που δεν έχουμε αρκετή πληροφόρηση για την ε, βιομάζα και την θνησιμότητα. Σε μια τέτοια αλία θεωρούμε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ανεπαρκούς τεκμηρίωσης αλία. Άρα δεν μπορούμε να δώσουμε επαρκείς συμβουλέ σε σχέση με τους στόχους διαχείρισης. Άρα είναι περιορισμένη η δυνατότητα διαχείρισης. Όμως είναι υπεραπλούστευση να θεωρήσουμε ότι τα αλλιεύματα χωρίζονται σε αυτές δύο κατηγορίες. Τα είδη. Υπάρχει μια μεγάλη κλιμάκωση ε, στην πληροφόρηση που έχουμε. Για ορισμένα είδη είμαστε πολύ κοντά στην ε, μία κατάσταση επάρκεια δηλαδή και πληθώρα στοιχείων, ενώ για κάποια άλλη, άλλα είδη δεν έχουμε σχεδόν καθόλου στοιχεία. Άρα δεν είναι άσπρο μαύρο η εικόνα. Γιατί δεν προσπαθούμε να έχουμε πληθώρα στοιχείων για όλα. Για τη συλλογή των στοιχείων και η επεξεργασία τους για να διατυπώσουμε μοντέλα και μετά συμβουλές ε, είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Άρα ίσως να μην έχει έννοια να θελήσουμε να έχουμε τέτοια πληθώρα για όλα τα είδη. Ίσως για κάποια από τα λιγότερες σημασία είδη θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι αρκούν μερικές γενικές αρχές διαχείρισης. Αν και για κάποια είδη δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να κάνουμε απευθείας αποτίμηση. Ακριβή αποτίμηση. Αρκεί να υπάρχουν ε, επαρκώς ρωμαλαίοι ε, κανόνες διαχείρισης. Λοιπόν, είναι πρόβλημα αυτές, ε, αυτά τα ίδια που δεν έχουμε υπαρκή στοιχεία για την Ευρώπη. Πρέπει να το εξετάσουμε πολύ. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, είδαμε τις συνολικές εκφορτώσεις όλων των ειδών στα ευρωπαϊκά λιμάνια. Στη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα, τον Βορειοανατολικό Ατλαντικό, τη Βαλτική και είδαμε τι ποσοστό αυτών των εκφορτώσεων και από πλευράς βάρους και από πλευράς αξίας ε, είναι από ήδη ε, με πληθώρα στοιχείων. Το εξετάσαμε ανά ετών και έχουμε εδώ στην έκθεση αναλυτική ε, παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Για το βάρος, στο Νοτιοανατολικό Ατλαντικό και την Βαλτική, όπου οι συμβουλές δίνονται από το Διεθνές Συμβούλιο για την εκμετάλλευση των θαλασσών, το 50% και για βάρος και για αξία είναι από είδη που θεωρούνται ανεπαρκούς τεκμηρίωσης. Στη Μεσόγειο και τον Εύξηνο ένα μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 80% των εκφορτώσεων είναι από είδη ανεπαρκούς τεκμηρίωσης. Και για τις δύο ομάδες περιοχών έχουν υπάρξει κάποιες αλλαγές το 2011. Η εκτίμησή μας ε, βασίζεται σε στοιχεία που υπέβαλαν τα κράτη-μέλη στο ΣΤΕΦΚ και κάποια κράτη δεν έστειλαν στοιχεία του 2011. Τώρα αυτό είναι συγκυριακό. Θα το δούμε περαιτέρω. Γενικά όμως αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Αλίας αφορά είδη για το οποίο δεν έχουμε παρκή στοιχεία. Εδώ έχουμε μια κατανομή ανά περιοχές. Εδώ είναι οι περιοχές ανάλογα και με τα συμβουλευτικά συμβούλια, τα περιφερειακά. Και με βάση, με, με τα βλητή αναφοράς, ε, το ευρώ. Βλέπετε ότι το μπλε τμήμα των πιτών είναι για τα ανεπαρκή είδη. Βλέπετε στη Βαλτική το, μεγαλύτερο, το μικρότερο τμήμα Το μεγαλύτερο τμήμα είναι από επαρκώς τεκμηρωμένα είδη, ενώ στον Εύξηνο όλα είναι από ανεπαρκώς τεκμηρωμένα. Στη Βαλτική όμως μόνο τρία είδη είναι πλήρως αποτιμημένα. Ενώ στη Μαύρη Θάλασσα έχουμε μεν 18 είδη που είναι πλήρως τεκμηριωμένα, αλλά έχουμε πολύ περισσότερα είδη. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλο το ποσοστό όπου χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Στη Βαλτική είναι πολύ απλούστερη η κατάσταση, πολύ πιο περιορισμένος αριθμός ειδών. Όπως σας είπα, τα ποσοστά εκφορτώσεων από τα μεν και τα δε είδη καλύπτονται πιο αναλυτικά και λυπάμαι γιατί στα τυπωμένα αντίτυπα δεν φαίνονται τα χρώματα. Τα μικρά σκάφη από, που είναι λιγότερο από 12 μέτρα μήκος ψαρεύουν περισσότερα ε, ανεπαρκώς τεκμηρωμένα είδη ενώ τα πελαγικά είδη αποτιμώνται καλύτερα ενώ τα σπόνδυλα όπως οι αστακοί, οι γαρίδες, τα καβούρια επίσης δεν καλύπτονται αρκετά. Και επίσης τα βαθυπελαγικά είδη δεν καλύπτονται επαρκώς. Ένα σημαντικό τμήμα λοιπόν των αλλιευμάτων μας δεν είναι επαρκώς τεκμηριωμένα. Γιατί? μία πλήρης αποτίμηση με βάση την ηλικία που είναι ο χρυσός κανόνας για την καλή αποτίμηση σημαίνει πληροφορίες για μια σειρά από στοιχεία εκφορτώσεις, απορρίψεις ανα ε, κατηγορία ηλικίας θέλουμε στοιχεία για τις τάσεις ε, βιολογική πληροφόρηση, πληροφόρηση για την θνησιμότητα την ηλικία ορίμανσης. Όταν έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να γίνει και περαιτέρω δουλειά για να φτιάξουμε ένα μοντέλο δυναμικής εκτίμησης του πληθυσμού για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε αποτιμήσεις σε σχέση με, τις, ε, με τους στόχους διαχείρισης. Δεν επιχειρήσαμε πλήρη ανάλυση όλων των ανεπαρκώς τεκμηρωμένων ειδών. Εξετάσαμε τα βορειοδυτικά ύδατα και από τα 20 πιο αλλιευόμενα είδη προσπαθήσαμε να καταλάβουμε γιατί κάποια από αυτά δεν είναι παρκώς τεκμηριωμένα. Και συνοπτικά υπήρχαν ε, περιορισμοί για όλα τα τέσσερα σημεία που προανέφερα. Δεν είχαμε αρκετή, ε, ε, αρκετά στοιχεία για τις απορρίψεις, δεν είχαμε ιδίως για τα ασπόνδυλα αρκετές ε, μελέτες για, την, ε, για το, το πόσο πολυπληθή είναι. Δεν είχαμε στοιχεία για το ρυθμό αύξησης και σε άλλες περιπτώσεις είχαμε όλα αυτά τα στοιχεία αλλά δεν είχαν εκπονηθεί μοντέλα. Δεν υπήρχε αρκετό ενδιαφέρον, δεν υπήρχε αρκετό προσωπικό για να κάνει τα μοντέλα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η ανεπάρκεια των στοιχείων που οδηγούν στην ανεπάρκεια τεκμηρίωσης. Αλλά υπάρχουν κενά στη διαδικασία συλλογής και αποτίμησης της ε, πληροφόρησης. Επόμενο θέμα. Από τα υποτεκμηριωμένα αυτά είδη, που είναι αρκετά, για πολλούς και διάφορους λόγους πώς γίνεται η αξιολόγηση και η διαχείρισή τους ευρωπαϊκά χωρικά ύδατα. Εδώ ισχύουν διαφορετικές προσεγγίσεις ε, στις ζώνες ΝΕΑΦΚΑ, Βαλτικής, ε, το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης των Θαλασσών δίνει συστάσεις και συμβουλές, ενώ για την Γενική Επιτροπή Αλίας της Μεσογείου καλύπτεται η Μεσόγειος και η Βαλτική θάλασσα. Όπως είπα και προηγουμένως, υπάρχει μια σχέση μεταξύ των μεθόδων αξιολόγησης των υποτεκμηριωμένων ειδών και των στόχων της ε, διαχείρισης. Δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση ε, με βάση μόνο κριτήρια μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, χωρίς ε, κάποιες οδηγίες για την διαχείριση ή κάποιες αναλλακτικές λύσεις. Γι' αυτό και οι επιστήμονες δίνουν κάποιες κατευθυντήρες γραμμές για όσους διαχειρίζονται την αλία. Γι' αυτό θα πρέπει να δίνονται ε, ποσοτικοποιημένα επιστημονικά απορίσματα, ιδιαίτερα για τα ε, υποτεκμηριωμένα είδη. Και είχαμε και μία νέα προσέγγιση της ISIS ε, από το 2012. Ιδιαίτερα στις ζώνες Διεθνούς Συμβουλίου για την Εξερεύνηση των Θαλασσών έχουμε ε, περισσότερο ε, ευρωπαϊκές οικονομικές, ε, αποκλειστική κοινοτική διαχείριση σε σχέση με τη Μεσόγειο και τη Βαλτική που δεν υπάρχει αμυγός κοινοτική διαχείριση. Σε ό,τι αφορά το Γενικό Συμβούλιο Ελίας Μεσογείου, εκεί υπάρχουν περιορισμοί σε ό,τι αφορά τα στοιχεία και τους πόρους. Δηλαδή δεν χρησιμοποιούνται όλα τα στοιχεία εξαιτία της έλλειψης των πόρων. Και η Επιστημονική Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή προσπαθεί να παράσχει τεχνογνωσία και πόρους και μάλιστα ε, εφάρμοσε κάποιε ε, μεθόδους ε, για υποτεκμηριωμένα είδη προκειμένου να προβεί σε κάποιες, έστω και μερικές αξιολογήσεις. Και μάλιστα βλέπετε στην παρένθεση τι εννοείται ως μέθοδος υποτεκμηριούμενο είδους. Αυτή τη στιγμή οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται για να δοθούν ποιοτικές συστάσεις διαχείρισης, χωρίς συστάσεις ποσοτικές. Σε ό,τι αφορά τη ζώνη του Διεθνού Συμβουλίου Εξερεύνησης Θαλασσών, έχουμε ε, περισσότερες μεθόδους αξιολόγηση υποτεκμηριωμένων ειδών. Δεν θα σας κουράσω με λεπτομέρειες, αλλά ξεκινώντας από την κορυφή προς τα κάτω, έχουμε διαφορετικά δεδομένα και μοντέλα που ε, εφαρμόζονται σε περίπτωση που έχουμε μόνο πληροφορίες για το αλίευμα και σε περίπτωση που έχουμε στοιχεία που μας επιτρέπουν μια πλήρη αξιολόγηση. Πάντως ε, έχουμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες ε, στις οποίες παρατηρείται ανεπάρκεια δεδομένων και εκεί δίνονται διαφορετικές συμβουλές. Για δεδομένα που αφορούν μόνο την αλίευση, που είναι πολύ περιορισμένα, δύσκολο είναι να δοθούν συμβουλές διαχείρισης μόνο κάποιες γενικές δηλώσεις μπορούν να γίνουν. Όταν έχουμε στοιχεία και για το, το αλίευμα και για την αυθονία του, μπορούν να δοθούν κάποιες συμβουλές με βάση τους στόχους της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Οπότε μπορούν να δοθούν κάποια στοιχεία, κάποιες συμβουλές για το κατά πόσο γίνεται βιώσιμη αλίευση κάποιων ε, ειδών και μπορούν να δίνονται επιστημονικές συμβουλές με βάση τις ευρείες αρχές της διαχείρισης, ακόμη και αν δεν έχει γίνει αξιολόγηση ως προς τους, ε, συγκεκριμέ... ως προς συγκεκριμένους στόχους της διαχείρισης. Τώρα, μοντέλα υπερπαραγωγής με περιορισμένα στοιχεία. Ε, μπορούν να δοθούν κάποιες συστάσεις με βάση τις ε, συνολικές αλλιεύσεις και τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, αλλά δυστυχώς οι συμβουλές αυτές είναι γενικού χαρακτήρα και δεν μπορούν να δοθούν ε, επιμέρους συμβουλές για συγκεκριμένους κανόνες ελέγχου, όπως είναι η διάσταση των διακαίνων των διχτυών και ούτω καθεξής. Σε άλλες αξιολογήσεις έχουμε πιο λεπτομεριακά στοιχεία για τον πληθυσμό των ψαριών ή την ανανέωση του πληθυσμού. Οπότε μπορούν να δοθούν κάποιες συμβουλές ό,τι αφορά τα υποκατάστατα ή την καταπροσέγγιση μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεν έχουμε τον ακριβή ορισμό της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης, αλλά θεωρούμε ότι έχουμε κάποια ε, ελάχιστη βιολογική γνώση για τη βιωσιμότητα του αλληλευτικού αποθέματος και με βάση αυτή την καταπροσέγγιση μέγιστη βιώσιμη απόδοση μπορούμε να δώσουμε κάποιες συμβουλές για τη διαχείριση. Πάντως ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε μια σταδιακή αύξηση της ροής των πληροφοριών όταν διαφορετικοί στόχοι διαχείρισης μπορούν να διευκρινιστούν για τα διάφορα επίπεδα διαθεσιμότητας των δεδομένων. Κάποιοι κανόνες κοινή λογικής εφαρμόζονται ώστε να εξασφαλίζεται βιώσιμη διαχείριση, ακόμη και αν αυτή δεν τηρεί πλήρως τους στόχους της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης. Αυτά για τη διαδικασία αξιολόγησης. Τώρα να σας αναλύσω τι χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν κάποιες αποφάσεις προς τη διαχείριση σε σχέση με υποτεκμηριωμένα αλληλευτικά είδη. Πριν το 2012, το Διεθνές Συμβούλιο δεν έδωσε ποσοτικές συμβουλές για υποτεκμηριωμένα είδη. Θεω... Απλώς μίλησαν για υπερεκμετάλλευση ή υποεκμετάλλευση και δεν έδωσαν συστάσει για συγκεκριμένα όρια μέγιστου του βιώσιμου συνολικού επιτρεπόμενου ελιεύματος, ΤΑΚ. Αλλά υπήρχε όλο και πιο ζωηρό ενδιαφέρον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ποσοτικέ επιστημονικέ συμβουλέ σε ό,τι αφορά τα όρια των ποσοστώσεων. Από το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε διάφορε δηλώσει ε, και εξέδωσε και χειρίδια πολιτική και διαχείριση με τους όρους για τη λήψη αποφάσεων για τα υποτεκμηριωμένα αυτά είδη. Εφάρμοσε περισσότερο όμως την κοινή λογική παρά επιστημονικά απορίσματα για να ορίσει τα, τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλλιεύματα και για πολλά χρόνια τα ΤΑΚ στηρίζονταν στο τεκμήριο ότι από τη στιγμή που υπήρχε ευθύνουσα πορεία ενός αλλιεύματος εφαρμόζονταν μείωση κατά 15% του ΤΑΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ενθάρρυνση, την πίεση της Κομισιόν προς, την, το Διεθνές Συμβούλιο να δίνει ποσοτικές ε, συμβουλές για τα ΤΑΚ σε σχέση με υποτεκμηριωμένα είδη, το 2012 το Διεθνές Συμβούλιο Εξερεύνησης ε, ε, Θαλασσών έδωσε μία προσέγγιση με ποσοτικές συμβουλές για μέγιστο επιτρεπόμενο, συνολικό επιτρεπόμενο αλίευμα σε υποτεκμηριωμένα είδη. Αυτό ισχύει φυσικά για τη ζώνη του Διεθνού Συμβουλίου και στηρίζεται στην αναγνώριση ότι μπορεί να έχουμε διάφορα επίπεδα γνώσης για τα αλληλευτικά αποθέματα. Δεν είναι άσπρο-μαύρο, δεν είναι δύο αμυγές κατηγορίες υποτεκμηριωμένα ή επαρκώς τεκμηριωμένα. Και επίσης καθορίστηκαν κάποιοι κανόνες διαχείρισης για διάφορες κατηγορίες δεδομένων. Για κάθε αλληλευτικό απόθεμα τα διαθέσιμα δεδομένα αξιολογούνται και τότε ε, περιλαμβάνονται τις κατηγορίες αξιολόγησης ανάλογα με τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα. Αυτό που απαιτείται είναι ένας συνδυασμός ε, των κανόνων διαχείρισης ε, που θα ανταποκρίνονται στις μεθόδους αξιολόγησης. Και φυσικά θα πρέπει να βρεθούν αποδεκτοί στόχοι της διαχείρισης ε, που θα ευθυγραμμίζονται με τα διαθέσιμα στοιχεία αυτό είναι προτιμότερο από το να αποφεύγεται οποιαδήποτε αξιολόγηση λόγω έλλειψης στοιχείων. Και μάλιστα η ISIS με την προσέγγιση για τα υποτεκμηριωμένα είδη επέτρεψαν κάποιο επίπεδο αβεβαιότητας εφόσον είχαν περιορισμένα στοιχεία και το Διεθνές Συμβούλιο ε, χρησιμοποίησε και ένα προληπτικό κριτήριο, μια γενική ε, μείωση 25% σε περίπτωση που δεν είχε τηρηθεί ένα συγκεκριμένο κατόφλι. Τώρα βλέπετε πώς τα διάφορα λεφτικά είδη καταχωρούνται στις κατηγορίες αξιολόγησης. Και βλέπετε που έχουμε πλήρη αξιολόγηση, βάση στοιχείων απογραφής, που έχουμε αξιολόγηση βάση στοιχείων απόρριψης ή εκφορτώσεων. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία καταγράφονται σε διαφορετικές κατηγορίες και ισχύουν και διαφορετικοί έλεγχοι και μέθοδοι διαχείρισης. Τώρα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, για να σας το εξηγήσω. Ένα παράδειγμα που αφορά ένα αποθέμα σελαχιού στην Κελτική θάλασσα στα χωρικά ύδατα μεταξύ δηλαδή Ηνωμένου Βασιλείο και Ιρλανδίας. Και βλέπετε στα δεξιά ε, το δέντρο αυτών των αποφάσεων και το κίτρινο στοιχείο θεωρείται ε, απόφαση με βάση πληροφορίες μελέτης και ε, οι πληροφορίες με βάση αυτής μελέτης στηρίζονται σε, ε, αλήψη της προηγούμενης χρονιάς και ελαμβάνεται υπόψη και, ένα, και η μείωση του αποθέματος. Χρησιμοποιείται δηλαδή ανάλογα με το αν αυξάνεται ή μειώνεται το απόθεμα. Χρησιμοποιείται αυτός πολλαπλασιαστής ε, για να υπολογιστούν τα τάκ. Και μια και μιλούμε για υποτεκμηριωμένο είδο υπάρχει και ένα επιπλέον προληπτικό κριτήριο που εφαρμόζεται στον υπολογισμό και που προβλέπει 20% μείωση επιπλέον στο ΤΑΚ, στην σύσταση για ΤΑΚ, προκειμένου να ε, ληφθεί υπόψη η ανεπάρκεια των στοιχείων. Οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η σύσταση του ΤΑΚ θα πρέπει να είναι μόνο 64% της προηγούμενης σύστασης για ΤΑΚ, δηλαδή ισχύει 36% μείωση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα της εφαρμογής του κανόνα της κοινή λογικής, παρά την ανεπάρκεια των στοιχείων και της έλλειψης άμεσης αξιολόγησης ως προς τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, γιατί δεν είναι γνωστή η μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Δεν θα ήθελα να επιμείνω περισσότερο σε αυτό. Να μιλήσω λίγο για τις αξιολογήσεις ε, της στρατηγικής διαχείρισης. Και θα ήθελα να σας μιλήσω γι' αυτό γιατί στο παρελθόν λέγαμε ότι καθορίζουμε τους στόχους διαχείρισης και αν δεν συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε, δεν πρόκειται να δώσουμε επιστημονικές ε, συμβουλές. Αντί να έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που οι στόχοι διαχείρισης προσδιορίζουν τις συμβουλές που απαιτούνται, μία εναλλακτική λύση θα ήταν να δεχτούμε ότι έχουμε ανεπαρκείς γνώσεις ή περιορισμένα δεδομένα, αλλά παρόλα αυτά να φροντίσουμε οι αποφάσεις μας για τη διαχείριση να λαμβάνουν υπόψη και αυτή την αβεβαιότητα ε, παρά να προσπαθούν να, την ε, καταργήσουν από το σύστημα. Αυτό που δείχνουν τα στοιχεία για, την, για τις αξιολογίες στρατηγικής διαχείρισης είναι ότι έχουμε μια προσωμείωση του μοντέλου με τη δυναμική του, στο, του, και τον ε, αντίκτυπο της αλίας. Μετά στα δεξιά έχουμε προσωμείωση για την συλλογή δεδομένων και τη διαδικασία αξιολόγησης. Αλλά ε, λαμβάνουμε υπόψη της, ε, την ανεπάρκεια των στοιχείων και τη συμπεριλαμβάνουμε στις προτάσεις ε, για τη διαχείριση. Έτσι έχουμε και ατελείς συμβουλές διαχείρισης που επιτρέπει όμως το διαχειριστικό μοντέλο να επηρεάσει το απόθεμα. Και έτσι λαμβάνουμε υπόψη την αύξηση, τη μείωση, τη σταθερότητα του ελευτικού αποθέματος. Αλλά τουλάχιστον έχουμε μια ρεαλιστική αποτίμηση και αναγνώριση της ανεπαρκούς γνώσης που έχουμε. Δεν μπορούμε να έχουμε τέλειες πληροφορίες και να γνωρίζουμε την ακριβή κατάσταση του αλληλευτικού αποθέματος και να κάνουμε και τέλειες προσομοιώσεις. Μπορούμε όμως να συγκρίνουμε διάφορους κανόνες αποφάσεων και να δούμε πώς ανταποκρίνονται σε αυτά τα ελευτικά αποθέματα. Και με προσομοιώσεις και με διαφορετικά επίπεδα σφάλματος καταλήγουμε σε παρατηρήσεις διαχείρισης και να αντικαταστήσουμε την έλλειψη στοιχείων μελετών από τις πολλαπλές αυτές προσωμιώσεις. Ή ε, κάνουμε προσωμιώσεις με, διαφορετικά, με διαφορετικές υποθέσεις για το βιολογικά χαρακτηριστικά του αποθέματος, αν δεν έχουμε στοιχεία για την ορίμασή του. Οπότε ε, δοκιμάζουμε συγκεκριμένους ε, διαχειριστικούς κανόνες με βάση διαφορετικές υποθέσεις κάθε φορά και βλέπουμε αν λειτουργούν. Το αριστερό πάνελ δείχνει πώς ε, τροποποιείται η βιομάζα. Και στα δεξιά βλέπουμε πώς αλλάζει η απόδοση της αλίας. Και το μέσο σημείο δείχνει πώς ε, εφαρμόζεται το μοντέλο διαχείρισης. Και στην περίπτωση αυτή μπορούμε να δούμε αν ο, ο διαχειριστικός κανόνας οδήγησε σε βελτίωση, στη βιομάζα του ελευτικού αποθέματος ή όχι για να οδήγησε σε βελτίωση της απόδοσης. Η μαύρη γραμμή είναι η μέση απόδοση και η διακεκομένη γραμμή είναι τα διάφορα επίπεδα εμπιστοσύνης. Να σας δώσω άλλο ένα παράδειγμα εδώ είναι σχεδόν το ίδιο. Έχουμε τρεις διαφορετικές σειρές όπου μια τέτοια ανάλυση που γίνεται με διαφορετικές προϋποθέσεις για το κατά πόσο η μελέτη ή όχι έδινε ακριβή ε, εκτίμηση για την αυθονία των αποθεμάτων ή αν βασιζόταν σε υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση της αυθονίας των ε, στόκ. Και στις δύο περιπτώσεις βλέπουμε ότι το απόθεμα βελτιώνεται και φτάνει στους στόχους βιομάζας, αλλά στην κάτω περίπτωση το απόθεμα τελικά δεν βελτιώνεται ώστε να φτάσει στο στόχο. Υπάρχει ωστόσο κάποια βελτίωση σε σχέση με την κατάσταση status quo. Μπορεί λοιπόν να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι αν και κάποιος κανόνας διαχείρισης μπορεί να μην είναι βέβαιος, ε, για κάποια φάσμα προσδοκιών σε κάθε περίπτωση ο κανόνας διαχείρισης που ελέγχεται εδώ οδήγησε σε βελτίωση της κατάστασης. Υπάρχουν άλλα παραδείγματα όπου κάποιος κανόνας διαχείρισης ελέγχεται και σε κάποιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι το, το καταραίει τελείως οπότε καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτοί οι κανόνες διαχείρισης δεν, είναι, ε, δεν ευσταθούν. Προσπαθώ να σας δείξω ότι ακόμα και αν δεν έχουμε πλήρη, απόλυτες γνώσεις, τέλειες γνώσεις, μπορούμε να ελέγξουμε κανόνες διαχείρισης που θα ε, στηρίξουν τη βεβαιότητά μας ή θα την μειώσουν σε ένα επίπεδο που θα θέλαμε. Τώρα, αυτές οι διαδικασίες αξιολόγησης των, της διαχείρισης έχουν εφαρμοστεί για διάφορες μεθόδους ε, διεθνείς ώστε να κάνουμε δηλαδή τέτοιες ε, αξιολογήσεις ε, για τις διάφορες μεθόδους management του ISIS. Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη λοιπόν. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια αναθεώρηση κάποιων διεθνών προσεγγίσεων και σύντομα να σας πω ότι κάποια βασικά μηνύματα που προέκυψαν εδώ είναι καταρχήν στη Βόρεια Αμερική και στην Αυστραλία σε σχέση με τις ε, τα ελλειπή σε στοιχεία στόκ ε, λαμβάνουμε υπόψη μια διαφορετική ιεραρχία κατηγοριών δεδομένων, διαφορετικούς κανόνες διαχείρισης που εφαρμόζονται στα διάφορα επίπεδα δεδομένων ώστε να μην μεταχειριζόμαστε τα στόκ ε, ως μαύρο ή άσπρο αλλά να έχουμε μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση με βάση τα δεδομένα που έχουμε και ανάλογα με την κατηγορία δεδομένων με την οποία ασχολούμαστε. Βέβαια υπάρχει πάντοτε η επιθυμία να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει διαρκώς μεγαλύτερη προφύλαξη όσον αφορά τους κανόνες ελέγχου της ε, διαχείρισης ε, και όσον αφορά την μείωση της βεβαιότητας. Όσο, περισσότερο, όσο λιγότερα στοιχεία υπάρχουν, τόσο μεγαλύτερη ε, προσοχή πρέπει να δίνεται στον έλεγχο τη διαχείρισης. Είναι το πιο ισχυρό αυτό εργαλείο για να αξιολογήσουμε πώς αποτελεσματικές είναι οι αποφάσεις διαχείρισης ενώπιον της αβεβαιότητας. Σε βάση περιπτώσει είναι μια διαδικασία υποεξέλιξη. Σε κανένα τομέα δεν έχουμε φτιάξει μια καθολική ε, μελέτη ή αξιολόγηση όλων των ε, τρόπων διαχείρισης με βάση ελληπή στοιχεία. Έχουμε όλοι να κάνουμε παγκοσμίω με μεθόδους και ανάπτυξη μεθόδων ε, σε σχέση με στόκο, με λυπή στοιχεία. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι στην Αυστραλία κάνουν πολύ ρητές δηλώσεις σε σχέση με την απέτηση όσον αφορά την ε, σχέση κόστος ωφέλειας για τη διαχείριση για μικρά αλλιεύματα δεν είναι, δεν ωφελεί από άποψη κόστος να προσπαθούμε να φτιάξουμε ε, ε, αποθέματα στοιχείων, μάλλον στοιχεία για τα αποθέματα και, να, και, και λένε ότι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους γενικούς κανόνες για να τα διαχειριστούμε αυτά γιατί δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στο να κάνουμε ακριβείς αξιολογήσεις για ένα μικρό απόθεμα για ένα μικρό αλλιεύμα. Τώρα, αν δούμε προς το μέλλον, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν και είπα εξ αρχή ότι αυτή η μελέτη καθαρά αφορούσε την αξιολόγηση των αποθεμάτων και όχι την ευρύτερη ανάγκη για πληροφορίες για τη διαχείριση των αλλιευμάτων, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι με την μεγαλύτερη εισαγωγή περιβαλλοντικών στόχων στη διαχείριση των αλλιευμάτων, η επιθυμία για επιβολή απαγορεύσεων, απορρίψεων κτλ., Αυτά τα προγράμματα για τη διαχείριση των αλλιευμάτων και η επιθυμία για καλύτερη διαχείριση θα αυξηθεί, πράγμα που έχει επιπτώσεις για τους πόρους που υπάρχουν για να αξιολόγηση των αποθεμάτων στην πιο κλασική περίπτωση διαχείρισης αλλιευμάτων. Και με το οικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρώπη επίσης φαίνεται να είναι αναπόφευκτο να δεχτούμε ότι χρειάζεται πως χρειάζεται να πετύχουμε και αξιολογήσεις όπου η αναλογία κόστος ωφέλειας να, είναι, να στέκει και αυτός, ε, αυτή, αυτός ο προβληματισμός θα ελέγχεται περισσότερο στο μέλλον. Σε σχέση με τα αλλιεύματα λοιπόν με λυπή στοιχεία υπάρχει μια αναλογία ευρωπαϊκών αλλιευμάτων που ε, θεωρείται ελλειπής. Και προφανώς αυτό είναι πρόβλημα. Σε πολλές περιπτώσεις ο κίνδυνο υπεραλίευσης δεν είναι ο ίδιο για όλα τα αποθέματα. Η συμπεριφορά πολλών από τους στόλους είναι, κατευθύνεται προς τα πιο πολύτιμα ή τα πιο εγκαταλειμμένα αποθέματα και οι αλλιευτικές ευκαιρίες καθορίζουν τον, τη συμπεριφορά του στόλου. Άρα λοιπόν τα αποθέματα που είναι λιγότερο ευάλωτα από τα βασικά εμπορικά είδη ή τα λιγότερα εκτεθειμένα αλλιεύματα από ότι τα κύρια εμπορικά μπορεί να μην κινδυνεύουν από υπεραλίευση από τη στιγμή που υπάρχουν ευκαιρίες για τα βασικά στόκο και διατηρούνται σε ένα επίπεδο ε, σταθερό και αντίστοιχο με την, με την μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ίσως όμως να μην είναι πρόβλημα λοιπόν το να μην έχουμε ε, ε, πλήρη στοιχεία για όλα τα αποθέματα. Μπορεί να είναι δυνατόν στρατηγικά να ορίσουμε κάποια βασικά αποθέματα επί τη βάση αυτών που καθορίζουν τη συμπεριφορά των αλληγμάτων ή των αποθεμάτων που είναι πιο ευάλωτα στον αντίκτυπο από την αλληλεία και σε σχέση με αυτά να μπορέσουμε να ορίσουμε τα όρια μέγιστης ε, βιώσιμης απόδοσης και ε, να την ορίσουμε και για τα υπόλοιπα είδη. Θα ήταν δηλαδή δυνατόν να έχουμε μια απλοποιημένη προσέγγιση παρακολούθησης και αξιολόγησης για κάποια από αυτά τα δευτερεύοντα αποθέματα και έτσι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν κάποιοι αυστηροί κανόνες ελέγχου ε, όσον αφορά την ε, αλίευση των συγκεκριμένων αποθεμάτων ενώ θα έχουμε πιο λεπτομερή στοιχεία για τα είδη τα οποία θεωρούμε πως είναι πιο ευάλωτα λόγω της μεγαλύτερης έκθεσης στην εκμετάλλευση συστάσει λοιπόν που προέκυψαν από αυτήν τη μελέτη, η πρώτη είναι να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση προ τι απαιτήσει συλλογή δεδομένων. Εδώ δεν επέμεινα. Όταν εξετάσαμε το συγκεκριμένο σημείο στη μελέτη, διαπιστώσαμε ότι κανένα κράτο μέλο δεν συμμορφούται απόλυτα προ τι απαιτήσει συλλογή στοιχείων με βάση το πλαίσιο συλλογή δεδομένων και στι περισσότερε περιπτώσει θα μπορούσαν να υπάρχουν βελτιώσεις στην ε, παροχή των στοιχείων. και στην παροχή των στοιχείων προς τις ε, ομάδες αξιολόγησης των στοιχείων. Θα είχαμε έτσι και καλύτερα αποτελέσματα. Με βάση τις ισχύουσες πάντα διατάξεις περί συλλογής στοιχείων. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν τέτοιες διατάξεις, καλό θα ήταν να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση προς αυτές. Όμως πέρα από αυτό, αν κανείς σκεφτεί λίγο πιο ριζοσπαστικά, Εάν ε, εξετάσει τα αποθέματα που αξιολογούνται αυτή τη στιγμή, έχουν εξελιχθεί τα πράγματα ε, διαχρονικά επί ad hoc βάσης, με βάση τα εμπορικώ σημαντικά στόκ ή τα αποθέματα από των οποίων υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Θα ήταν ίσως λοιπόν σωστό να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να διεξάγουμε μια στρατηγική ιεράρχηση των αποθεμάτων σε σχέση με τα επιθυμητά επίπεδα πληροφόρησης που χρειαζόμαστε και αυτά και να ορίσουμε έτσι ένα σύνολο ε, δεδομένων ή μεθόδων αξιολόγησης που είναι αποδεκτές για τα πιο ευάλωτα αποθέματα, ενώ για τα μικρότερα δευτερεύοντα είδη να πούμε συγκεκριμένα ότι δεν θα προσπαθήσουμε καν να φτάσουμε σε όλα αυτά τα στοιχεία, διότι πιστεύουμε ότι από τη στιγμή που τα κύρια αλλιεύματα, κύρια αποθέματα τα διαχειριζόμαστε σε σχέση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση, σημαίνει πως και τα υπόλοιπα στόκ θα είναι πιο στεναρά Methods are suggested. It's important to evaluate the practical implications. Όταν εξετάζονται νέες μέθοδοι για την πρακτική εφαρμογή αυτών των διαδικασιών, θα ήταν δυνατόν να μπορέσουμε να προβλέψουμε για ένα μειούμενο στόκ σημαίνει ότι αν δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για ένα συγκεκριμένο στόκ, μπορεί να υπάρξει και λιγότερη μείωση στη διαθέσιμη απόδοση. Οπότε οποιαδήποτε διαστρωματική προσέγγιση στη, στο, στη, στην αξιολόγηση των αποθεμάτων δεν θα οδηγήσει σε αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την παροχή πληροφοριών. Επίσης θα πρέπει να έχουμε και όρια κινδύνου ώστε οι επιστήμονες να μπορούν να θεσπίζουν διάφορες διαδικασίες σε σχέση με αυτά τα όρια έτσι και θα υπάρχει και ένας αμοιβαίος διάλογος και συνεννόηση για το ποια στοιχεία μπορούν όντως να δοθούν και ποια είναι τα αποδεκτά υποκατάστατα για τη βιώσιμη διαχείριση. Τέλος, όταν εξετάζουμε μελλοντικές δράσεις σε σχέση με τις, ε, τα, ελληπή, μάλλον, τα αλλιεύματα με ελληπή στοιχεία, θα πρέπει καλύτερα να εξασφαλίσουμε πως οι στόχοι της διαχείρισης είναι συνεπείς με τους πόρους που υπάρχουν για την ε, ε, παροχή αξιολόγησης και συμβουλή για τη διαχείριση. Γιατί διαφορετικά μπορεί να σχεδιαστεί ένα σύστημα το οποίο να μην μπορεί να σταθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την αναλυτική πληροφόρηση. Να αρχίσουμε τώρα ένα γύρο με τους βουλευτές. Που ζητάνε το λόγο. Ο κύριος Στίβενσον. Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Όταν μιλήσατε για αυτό που είπατε ότι εάν μειώνει το αριθμό των στοιχείων τότε χρειάζεται περισσότερη προληπτική δράση. Εμείς είχαμε πει ότι στο βόρειο-ανατολικό Ατλαντικό εάν για κάποια είδη δεν είχαμε αρκετά στοιχεία, μειώναμε κατά 10% το τάκ το χρόνο. Και οι αλλοί μου έλεγαν ότι ναι, δεν είχαμε στοιχεία, αλλά υπήρχε μεγάλος αριθμός και απλώς αυξάνονταν οι απορρίψεις με τον τρόπο αυτό. Νομίζω αυτό είναι αντιφατικό σε σχέση με την προσπάθειά μας δηλαδή να μειώσουμε τις απορρίψεις. Βεβαίως η αρχή της πρόληψης ε, είναι λίγο υπερβολικά χοντρικό όργανο. Υπερβολικά αμβλή. Οξύνει το πρόβλημα που προσπαθούμε να επιλύσουμε. Ποια είναι η γνώμη σας. Η κυρία Λόβιν. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Όλες σας οι συστάσεις ε, μου φαίνονται πολύ καλές. Ελπίζω και η Κομισιόν να τις λάβει υπόψη. Ερώτηση. Μιλήσατε για κόστος, ε, σχέση κόστους αποτελεσματικότητας. Μπορείτε να μας κάνετε μια εκτίμηση. Τι στοιχίζει η εκπόνηση ενός ε, μοντέλου πληθυσμού για κάποιο είδος. Μας είπατε ότι έχετε τα στοιχεία για, κάποια, για κάποιο είδος, αλλά δεν έχετε μοντέλο. Μπορείτε παρακαλώ να μας πείτε πόσο στοιχίζει. Πόσο κοστίζει η δουλειά που πρέπει να γίνει. Συμφωνώ με την νέα κοινή αλληλευτική πολιτική που είναι πιο φιλόδοξη. Η πιο φιλόδοξη που έχουμε ποτέ ψηφίσει ως Επιτροπή. Άρα θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερα δεδομένα για τα διάφορα είδη. Είναι σκανδαλώδες. 80% του βάρους ε, των ε, εκφορτώσεων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα να είναι υποτεκμηριωμένα ήδη και 50% στις άλλες θάλασσες. Μιλήσατε για το βάρος, αλλά όχι για τον αριθμό ειδών. Μήπως μπορείτε να μας πείτε πόσα είδη τον αριθμό των ειδών όπου δεν έχουμε επαρκή στοιχεία και όχι να μας μιλήσετε για το βάρος των εκφορτώσεών τους. Επίσης, οι συστάσεις σας. Βλέπω ότι προτείνεται ένα κατάλογο στρατηγικών προτεραιοτήτων που είπατε ότι θα έπρεπε να είναι τα είδη που αλλιεύονται κυρίως ή τα πιο ευάλωτα. Στόχος μας πρέπει να είναι πάντα να μην υπεραλλιεύσουμε τα πιο ευάλωτα είδη, γιατί κινδυνεύουν να εξαφανιστούν τότε. Αυτή θα έπρεπε να είναι η προτεραιότητά μας σε οποιαδήποτε μεικτή αλία. Έτσι για παράδειγμα αλλιεύουν στις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι βεβαίω πιο πολύ εκτίμηση αυτό από πλευρά μου. Ίσως όμως θα ήθελα και τη δική σας γνώμη. Πόσα υποτεκμηριωμένα ευάλωτα είδη έχουμε. Βεβαίως, οι διαχειριστικές πρακτικές δεν θα πρέπει να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες μειώσεις της χωρίσης στοιχείων. Δεν θέλουμε ε, να μην μας δίνουν στοιχεία οι αλληλείς για να μην υπάρχουν πιο αυστηροί κανόνες. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Είπατε ότι ορισμένοι δεν παρέχουν τα στοιχεία που υποχρεούνται. Δεν θα πρέπει να επιδείξουμε καμιά ανοχή για τέτοια παρακόλληση. Και στα πλαίσια της νέας αλληλευτικής, της νέας πολιτικής μας είπατε ότι κάποια στοιχεία μπορεί να μην αξιοποιούνται. Αλλά ότι πολλοί δεν συμμορφούνται με το πλαίσιο συλλογής στοιχείων. Τέλος, οι συστάσεις σας είναι ότι πρέπει να καθορίσουμε το αποδεκτό κατόφλι κινδύνου για τις ε, διαχειριστικές μας πρακτικές. Θα μπορούσα να συμφωνήσω. Αλλά εσείς ως επιστήμον μπορεί να έχετε αυτή την άποψη. Αλλά εμείς είμαστε πολιτικοί. Εκλεγόμεθα. Πρέπει εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη αυτού του κινδύνου. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μεγάλη διαφάνεια Πλήρε διαφάνεια για το πώ γίνεται αποτίμηση των αποθεμάτων, ιδίω όσον αφορά τα υποτεκμηριωμένα είδη, τη μεικτή αλληλεία. Με ανησυχεί λοιπόν κάπω κάποια ασάφεια για τον τρόπο εκτίμησης των αποθεμάτων για τα υποτεκμηριωμένα είδη. είναι απαραίτητη η διαφάνεια για το πώς γίνονται αυτές οι εκτιμήσεις. Γιατί αλλιώ μπορεί να αυξηθούν οι πιέσεις από πλευρά των διαχειριστών προς τους επιστήμονες να τους δώσουν κάποια στοιχεία. Και το είπατε στην παρουσίασή σας. Είπατε, μα ζητάνε πραγματιστικές συμβουλές. Άρα μπορεί να σας φέρει σε δύσκολη θέση. Και η τελευταία, η σας σύσταση είναι άρεστη. Πρέπει να διασφαλίσουμε συνέπεια μεταξύ πολιτικών στόχων και πόρων. Πρέπει να έχουμε τα στοιχεία τα κράτη-μέλη. Πρέπει να έχουμε τους αναγκαίους πόρους, ούτως ώστε οι οργανισμοί, ISIS, TEFC, να μας δίνουν την πληροφόρηση που θέλουμε για να καταλήγουμε σε υπεύθυνες αποφάσεις διαχείρισης των αποθεμάτων. Πολλά είπα, αλλά είναι μεγάλο το θέμα, γιατί είναι μεγάλο το ποσοστό των υποτεκμηριωμένων αλλιευμάτων. Είναι τεράστια πρόκληση όλα αυτά. Πρέπει να πάρουμε υπεύθυνε αποφάσεις για όλα αυτά τα αποθέματα. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μελέτη, την παρουσίαση και ελπίζω ότι θα αντιμετωπίσουμε με υπεύθυνο τρόπο τα θέματα αυτά και να ακούσουμε και την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Λοβίν. Δεν υπήρχαν άλλες ερωτήσεις. Να δώσω το λόγο στους ε, εκπονητές της μελέτης. Ο κύριος Δεγκάν. Για τα σχόλια του κυρίου Στίβενσον η αρχή της πρόληψης που είναι σε αυτή την προσέγγιση του ISS το 20%, 20% όχι 10%, 20% μείωση. Είναι μία μοναδική, δεν είναι αιτήσια μείωση. 10% ανά έτος θα δημιουργήσει απορρίψεις. Μία 20% μείωση από το ISIS μία και έξω για μια σειρά ετών σημαίνει ότι έχουμε μια σειρά ετών για να δούμε πώς θα αντιδράσει το είδος. Μειώνοντας λοιπόν την ε, αλλιευτική προσπάθεια θα πρέπει να μετρήσουμε την αντίδραση του αποθέματος για να δούμε εάν η συγκεκριμένη ποσόστοση είναι πλέον ε, βιώσιμη. Χρειαζόμαστε 5-10 χρόνια ένα περιθώριο για να δούμε βιολογικά τεκμηριωμένη, δηλαδή να έχει βιολογική έννοια ε, η μεταβολή του αποθέματος. Το θέμα των απορρίψεων. Θα εξαφανιστεί από τη μεταρρύθμιση της ΚΑΛΠ γιατί υπάρχουν υποχρεώσεις εκφόρτωσης. Αυτά τα δύο μέτρα από μαζί θα βελτιώσουν αυτή την κατάσταση. Ούτω ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμα τα ίδια αυτά με βάση τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Για το κόστος ε, του πλαισίου συλλογής στοιχείων υπάρχει ένα στοιχείο στη σελίδα 31 που δείχνει πόσο συμμορφούνται με τις υποχρεώσεις τους αυτές τα κράτη. Δεν έχουμε στοιχεία για ποσά, αλλά η ομάδα που αποτιμάει την συμμόρφωση εξετάζει και το κόστος. Σίγουρα θα υπάρχει μια έκθεση του STCF που θα περιέχει ε, αριθμητικά ποσά, αλλά δεν τα έχουμε τα στοιχεία αυτά. Εμείς. Δεν είναι απλός υπολογισμός αλλά πρέπει να γίνει. Πόσα είδη και όχι το βάρος. Απλώς. Είτε έχουμε επαρκή στοιχεία είτε όχι. Με βάση το πλαίσιο του ICs το ISIS δίνουν συμβουλές για περίπου 200 είδη, εκ των οποίων 122, δηλαδή 60-70% είναι υποτεκμηριωμένα. Μεγάλο ποσοστό. Για το κατόφλιο ε, κινδύνου. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για την ε, διαφάνεια. Αυτά τα κατόφλια πρέπει να τα δούμε στα πλαίσια συνολικά του συστήματος διαχείρισης. Είναι εύκολο να πούμε ποιο είναι ο κίνδυνος ε, η ε, θνησιμότητα να αυξηθεί ή να μειωθεί το απόθεμα. Πρέπει να δούμε συνολικά το κόστος όμως και το, συνολικά συγγνώμη τον κίνδυνο. Δεν μπορούμε να εξετάσουμε μόνο μία παράμετρο του συστήματος διαχείριση. Πρέπει να αποτιμήσουμε από κοινού όλους τους λόγους αβεβαιότητας. Δεν ξέρω αν έχει να προσθέσει τίποτα συντομία για το κατά πόσο θα πρέπει να επικεντρώσουμε τους πόρους ε, στα πιο ευάλωτα είδη σε σχέση με τα πιο ε, αλλιευόμενα. Το θέμα είναι ότι οι αλλιευτικές εργασίες ε, στοχεύουν σε συγκεκριμένα αλλιευτικά είδη. Και ανάλογα με το που ψαρεύουν και με τι αλληλευτικά εργαλεία αλλιεύουν, ε, ε, προσβλέπουν σε ένα μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα. Και φυσικά τα πιο εκτεθειμένα στην αλλιεύση ήδη είναι αυτά που υπόκειται και τις περισσότερες επιπτώσεις. Οπότε, σε ό,τι αφορά την ευπάθεια, το θέμα είναι πρώτον πόσο ευαίσθητο ευπαθέ είναι απέναντι στη θνησιμότητα το συγκεκριμένο αλλιευτικό είδο και πόσο εκτεθειμένο είναι στη θνησιμότητα το συγκεκριμένο είδο. Και σίγουρα τα πιο ευπαθή είδη είναι αυτά που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη θνησιμότητα. Ενώ μπορεί να είναι πιο ευαίσθητα κάποια αλλιευτικά είδη, αλλά ακριβώ επειδή δεν υπεραλλιεύονται, ιδιαίτερα δεν είναι και τόσο ευάλωτα. Οπότε θα πρέπει να δοθεί μια στρατηγική προσέγγιση και να γίνει διάκριση μεταξύ των ε, πιο αλλιευμένων ειδών και των πιο ευαίσθητων ή πιο ευάλωτων, ανάλογα με το πόσο εκτεθειμένα είναι. Πάντως η ευπάθεια στην ε, υπεραλήψη είναι σημαντικός παράγοντας. Και τώρα, ε, σε ό,τι αφορά τα ευπαθή ελευθερικά αποθέματα και τα περισσότερα είναι υποτεκμηριωμένα. Οπότε είναι και πιο εκτεθειμένα στη θνησιμότητα. Και τα ευαίσθητα από βιολογική άποψη ελευθερικά αποθέματα δυστυχώς σε, σε μεγάλο βαθμό είναι υποτεκμηριωμένα. Καταρχήν, τι εννοούμε υποτεκμηρίωση σε αυτή τη μελέτη για τα λευτικά αποθέματα. Λαμβάνοντα υπόψη και τι εκτιμήσει βιομάζας και την θνησιμότητα σε σύγκριση με του στόχου μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Γίνονται έρευνε και υπάρχουν πληροφορίε, οπότε δεν υπάρχει κενό δεδομένο σε ό,τι αφορά του στόχου τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Ελπίζω να απαντήθηκαν οι απορίε σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά για το έργο σας, για τη μελέτη σας, την παρουσίαση και σας απαλλάσσουμε. Α, συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει το λόγο και το ξέχασα. Καλησπέρα σας. Δεν είναι τη Σόνη και καλά θέλαμε το λόγο, αλλά σκόπιμο θα ήταν να κάνουμε κάποια σχόλια και να συμπληρώσουμε τη συζήτηση. Καταρχήν, να συγχαρώ τους κυρίους Λεκέν και ο Μπράιαν για την ε, εξαιρετική τους και πολύ τεκμηριωμένη έκθεση που μας ε, κάνουν, κάνει μια πολύ επίκαιρη και μεστή επισκόπηση ε, σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των στοιχείων για τα λευτικά είδη. Περιεκτική έκθεση, παραλαμβάνω, ενημερωμένη και επίκαιρη, γιατί λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της νέας προσέγγισης που ζητήσαμε από την ISIS και που άρχισε να εφαρμόζεται από το 2012. Οπότε από αυτή την άποψη η έκθεση και ως προς το περιεχόμενο και την ανάλυση, αλλά και ως προς τις συστάσεις της, είναι χρήσιμη στη συζήτηση. Λίγα σχόλια. Να μην υποτιμούμε το εύρος και την περιπλοκότητα του θέματος των δεδομένων. Τα δεδομένα δεν αφορούν μόνο την αλίευση, αλλά και την αλευτική προσπάθεια και τα δραστηριότητες του αλευτικού στόλου. Πρόκειται για ένα ε, ευρύ φάσμα στοιχείων. Τα περισσότερα χορηγούνται από τους αλείς και μέσω των κρατών μελών στα επιστημονικά Ινστιτούτα. Όλη αυτή η ροή των δεδομένων είναι αρκετά δαπανηρή και μερικές φορές καλούμαστε να κάνουμε επιλογές, είτε ατομικές είτε συλλογικές. Σε ό,τι αφορά την κάλυψη, δεν πρόκειται να αφισβητήσω αυτά που είπε ο κύριος Λεκέν στην τελευταία του παρέμβαση, αλλά προσπαθούμε τουλάχιστον να αποφύγουμε ε, την υποτεκμηρίωση τουλάχιστον στα πιο ευαίσθητα ελευτικά αποθέματα. Τα βαθύβια είδη, για παράδειγμα, που όπου γίνεται η αλλιεύσή τους ε, τις τελευταίες δεκαετίες μόνο, εκεί όντως υπάρχει ένα κενό δεδομένων, αλλά σιγά σιγά συμπληρώνουμε τα κενά και ε, τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να προβούμε σε αξιολογήσεις των αλλιευτικών αποθεμάτων. Και αυτή είναι δύσκολη, η πιο δύσκολη περίπτωση, αλλά είχαμε αρκετά αποθέματα σε κακή κατάσταση και εκεί υπήρχε σε μεγάλη πρόοδο, ε, γιατί ενισχύθηκαν πολλοί οι προσπάθειές μας προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη με δεδομένα. Μπορεί δηλαδή να μην είχαμε από την αρχή ή να μην είχαμε πάντα μια συστηματική προσέγγιση για τα ποια αποθέματα να καλύψουμε και σε ποια να δώσουμε προτεραιότητα, αλλά στην πορεία έχουμε εξασφαλίσει κάλυψη και για τα πιο σημαντικά είδη και για τα πιο ευαίσθητα είδη, αλλά και τα πιο πολύτιμα από άποψη ε, αξίας, τιμής ή τα πιο απειλούμενα ή τα πιο ευρεία αποθέματα, Αυξήθηκε λοιπόν ο αριθμός των αποθεμάτων που καλύπτονται. Υπάρχει πρόοδος και προς τον όγκο και ως προς την αξία των καλυπτόμενων αλληλευτικών αποθεμάτων. Και όλο και ελαττώνεται ο αριθμός των υποτεκμηριωμένων ειδών. Έχουμε για παράδειγμα ένα, ένα απόθεμα με τάκ 75 ε, τόνους. Δεν είναι και ιδιαίτερα αξιόλογο ε, αλληλευτικό είδος, οπότε θα πρέπει να κάνουμε επιλογή. Αξίζει ε, να κάνουμε έξοδα για την συγκέντρωση στοιχείου για το συγκεκριμένο αλληλευτικό είδος που είναι τόσο μικρό. Είναι αποδοτική μια τέτοια επιλογή. Αυτή είναι μια ε, επιλογή διαχείριση. Τέτοιου είδους ε, επιλογές τις κάνουμε καθημερινά και μερικέ φορέ επιλέγουμε να μην επενδύσουμε περαιτέρω σε ένα συγκεκριμένο αλληλευτικό είδο. Τώρα, πέραν τη υποτεκμηρίωση κάποιων αλληλευτικών αποθεμάτων, να δούμε πώ θα χρησιμοποιήσουμε τις συστάσεις του Διεθνού Συμβουλίου εξερευνηση των Θαλασσών για να βελτιώσουμε τι ε, αποφάσει και τι συμβουλέ διαχείριση. Και η προσέγγιση για τα υποτεκμηριωμένα είδη είναι ένα βήμα πρόοδου, γιατί ε, απομακρυνόμαστε πλέον από τα αποθέματα για τα οποία δεν έχουμε καμία συμβουλή σε αποθέματα που έχουμε και ποιοτικέ ε, συστάσεις και ποσοτικές. Και μάλιστα στην ανακοίνωση για τις ελευτικές ε, ευκαιρίες που και δυνατότητες που δημοσιεύσαμε τον περαμένο μήνα βλέπετε την πρόοδο που έχουμε. Έχουμε βελτίωση κατά 30 ελευτικά είδη, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει όντως πρόοδος. Τώρα, είναι ανάγκη να γίνει κάποια αναθεώρηση της κατανομής των πόρων. Γιατί λίγα είναι τα κονδύλια και για την ε, συλλογή των ε, δεδομένων και για τα επιστημονικά στοιχεία και γενικώ τους και στους ανθρώπινους πόρους έχουμε έλλειψη. Οπότε πρέπει να κάνουμε μια ορθολογική διαχείριση των πόρων προκειμένου να μπορέσουμε με αποτελεσματικότητα να χρησιμοποιήσουμε τα λίγα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα και να κάνουμε τεκμηριωμένε επιλογέ. Ποια θα είναι η βάση των μελλοντικών μα επιλογών. Και ίσω ο συνάδελφο θα δώσει κάποιε προτάσει για το τι με Ω προ τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΛΠ, έχουμε πια συμβουλές για περισσότερα λευτικά είδη, οπότε χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για τα αποθέματα, την αλληλεπίδραση μεταξύ των αποθεμάτων και τις ε, επιπτώσεις αυτής της αλληλεπίδρασης ε, εκεί που είχαμε αμυγή αλίευση έχουμε μεικτή αλίευση, δηλαδή αλίευση ταυτόχρονα πολλών αλιευτικών ε, ειδών και βλέπουμε και πώς αυτό το νέο στοιχείο επηρεάζει τις πολιτικές και οι επιλογές σε, μία, σε ένα αλιευτικό είδος επηρεάζουν ε, και τα άλλα αλιευτικά είδη, μια και γίνονται μεικτές αλιευτικές προσπάθειες. Επίσης έχουμε και την κάλυψη των, των σχεδίων που θα πρέπει οπωσδήποτε να στηρίζονται σε αδιάστα επιστημονικά κριτήρια και κάτι άλλο που αναφέρθηκε στη συζήτηση. Ε, χρειάζεται διάλογος με τους ενδιαφερόμενους, κυρίως με τον κλάδο, με τους ελίες, γιατί αυτοί προσδιορίζουν τις στρατηγικές αλλιεύσεις. Γι' αυτό και χρειάζονται τις γνώσεις και τις αξιολογήσεις. Και σε λίγα χρόνια καταφέραμε να έχουμε μέγιστη βιώσιμη απόδοση για όλα τα ελευτικά είδη. Τώρα χρειαζόμαστε και τις τιμές που θα καθορίζουν την μέγιστη βιώσιμη απόδοση και τη σχετική στρατηγική. Αυτές είναι οι βασικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτικής. Και μία παρατήρηση επιπλέον σε σχέση με αυτά που είπε η κυρία Λέβεν. Είπε ότι είναι κάπως αδιαφανής η διαδικασία, κάπως σκοτεινή. Δεν ξέρω τι εννοεί, αλλά διαφωνώ. Εγώ θα έλεγα, δεν θα έλεγα ότι έχουμε την απόλυτη διαφάνεια, αλλά και ε, αυτό που είπατε ότι υπάρχει αδιαφάνεια είναι ανακριβές. Μπορεί να μην είναι κατανοητά όλα αυτά σε όλους τους κυρίους θυντούς, γιατί ακόμη και εγώ έχω μερικές φορές απορίες για τα μοντέλα, αλλά δεν νομίζω ότι ο όρος αδιαφανής χαρακτηρίζει αυτή τη διαδικασία. Ίσα ίσα είναι διαφανής η διαδικασία και η συλλογή και η διαθεσιμότητα των δεδομένων και όλες οι αξιολογήσεις ε, είναι προσιτές Οπότε θα έλεγα να αποφεύγουμε τέτοιους χαρακτηρισμούς αδιαφανής ή σκοτεινή διαδικασία. Και να δώσω το λόγο στον συνάδελφο που θα σχολιάσει την ειδική κατάσταση στη Μεσόγειο θα είμαι σύντομο, εδώ ονομάζομαι Ζιλονιάν, με σημείο επαφή ανάμεσα στην ε, Κομισιόν και το ISIS. Δύο λόγια για να σα πω πού βρισκόμαστε. Αλλά καταρχήν θα ήθελα να πω ε, ότι η πρώτη σύσταση τη έκθεση, η συμμόρφωση με τι απαιτήσει συλλογή στοιχείων είναι φυσικά πολύ σημαντική, διότι η εισαγωγή της προσέγγισης αυτής από το ISIS πέρυσι σημαίνει ότι είναι ένα τεράστιο βήμα και ότι κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων στοιχείων. Χρειαζόμαστε δηλαδή στοιχεία και που αυτό απαιτείται το ISIS, το και, τα... και εμείς θα πρέπει να τα έχουμε. Φυσικά αυτή η προσέγγιση είναι υπό εξέλιξη, που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα πέρσι, γιατί το 2012 το ISIS ανέλησε 84 αποθέματα με περιορισμένων στοιχείων και μπόρεσε να δώσει ποσοτικές συμβουλές για τα 68 από αυτά. Φέτος το ISIS θα ξανακινήσει και θα επανεξετάσει κάποιες από αυτές τις ε, συμβουλές και αυτός και θα αξιολογήσει άλλα νέα στόκ που θεωρούνται ε, ως ε, λοιπόν τεκμηριωμένα. Ζητήσαμε επίσης από το ISIS να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες ανά στόκ για όλα τα στόκ με λυπή τεκμηρίωση, όπως και παράδειγμα να δούμε ποια στοιχεία θα χρειάζονταν για να βελτιωθεί η κατάσταση και ποιες είναι οι αναμενόμενες προθεσμίες για να έχουμε ποσοτικές πληροφορίες. Τώρα, σε σχέση με τη διαφάνεια, να προσθέσω απλά ότι αυτό που ζητήσαμε από το ISIS όσον αφορά τα περιορισμένα στοιχεία στοιχείων μάλλον από θέματα είναι στο Μνημόνιο Συνεννόησης και είναι δημοσιευμένα στο site του ISIS. Επίσης η προσέγγιση αυτή αναπτύσσεται στο site του ISIS και έχουμε επίσης αποφασίσει να διοργανώσουμε ειδική κατάρτιση με, το, με εμπειρογνώμενους του ISIS Αυτά, αυτή η κατάρτιση είναι ανοιχτή για όλους όσους ενδιαφέρονται και η προσέγγιση περιορισμένων στοιχείων συζητείται εδώ. Σε σχέση με το ΜΕΝΤ, να πω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο συνεννόησης ανάμεσα στην ISIS ε, και την ICM. Ε, από όταν ξεκινά κατάρτιση για κάποιους από τους εμπειρογνώμονες για διάφορα θέματα ε, και φυσικά το θέμα των αποθεμάτων με περιορισμένα στοιχεία είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα. Ευχαριστώ. Bien, muchas gracias. Άλλος κανείς, θέλει κανείς να προσθέσει κάτι. Αλλά παρακαλώ, πολύ σύντομα. Όχι. Δεν θέλει, άλλος κανείς, θέλει άλλος κανείς το λόγο. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς συνεχίζουμε. Μου, μου λέει η γραμματεία ότι το σημείο 11 της ημερήσης διάταξης ε, ειδικέ δράσει στην κοινή ελευθερική πολιτική για την άφηση του ρόλου των γυναικών ε, περίσσεψε από την πρωινή ημερήσια διάταξη. Δεν είχαμε το χρόνο να το αναλύσουμε το πρωί, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να το καλύψουμε έστω και εν συντομία τώρα το απόγευμα. Α μην μακρηγορήσουμε όμω για να προλάβουμε να καλύψουμε και τα υπόλοιπα σημεία. Αν αρκεστείτε σε ένα δεκάλεπτο θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε την πρωινή συζήτηση. Μα δεν έγινε καν συζήτηση. Α, συγγνώμη, δεν κατάλαβα καλά. Νόμιζα ότι είχατε ξεκινήσει τη συζήτηση το πρωί. Η κυρία Καραβάγιο, συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε ξεκινήσει και απλώς έμεινε, έμειναν λίγες Και Κανένα πρόβλημα κύριε Πρόεδρε. Απλώς ξεπεράσαμε τη συζήτηση, ξεπεράσαμε το χρόνο μας γιατί αναπτύχθηκαν πολύ πιο εκτενώς τα προηγούμενα θέματα και δεν προλάβαμε να αναφέρομαι, να αναφερθούμε στο δικό μου. Εγώ έχω μια συνεδρία στις 6.30, γι' αυτό και δεν έχω και πολύ χρόνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλα τα μέλη της Επιτροπής Αλίας, γιατί χάρη στις δικές τους προτάσεις, το ενδιαφέρον τους, την εμπειρία τους και τα σχόλιά τους, κατάφερα να συγκεντρώσω πολλές ε, καλές ιδέες. Πριν από ένα χρόνο ανέλαβα ε, την ιδιότητα του τακτικού μέλους των ε, Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Αλληλευτική Επιτροπή και εκεί ε, μου είπαν ότι θα πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα της ισότητας των δύο φύλων και της ισότητας των ευκαιριών σε όλους τους κοινωνικούς τομείς. Στην περίπτωση αυτή μας ενδιαφέρει η συμμετοχή των γυναικών στην κοινή αλληλευτική πολιτική. Και μάλιστα εγώ ανέλαβα να συντονίσω τη διάσταση του φύλου σε όλες τις πολιτικές και να συγκεντρώνω τα σχετικά στοιχεία. Είμαι αρμόδια για το gender mainstreaming, όπως λέμε και στα αγγλικά. Και στην προσπάθεια αυτή συγκέντρωση όλων αυτών των στοιχείων είχα τη μεγάλη χαρά να γνωριστώ με πολλούς ευρωβουλευτές και να διαπιστώσω και το έργο που γίνεται και σε άλλες επιτροπές. Και μπορώ να σας πω ότι με ιδιαίτερη ικανοποίηση διαπιστώνω ότι είμαστε η μόνη επιτροπή που κάναμε το καθήκον μας και συγκεντρώσαμε σε ένα έγγραφο τα διάφορα σχόλια από εκθέσεις, από δημόσιες ακροάσεις που αφορούν το θέμα της ισότητας. Και σας ευχαριστώ θερμά για τις προσπάθειές σας, γιατί και συμβάλλατε σε αυτή την ε, συμπίληση. Είναι σημαντικό να έχουμε συνέχεια κατά να έχουμε κατά νου τη συμμετοχή των γυναικών στις διάφορες φάσεις ε, της ε, αλίας και το ρόλο τους ε, στην αλία. Γιατί πραγματικά προσφέρουν τα μάλα και από οικονομική και από κοινωνική άποψη, συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του αλληλευτικού κλάδου και την περιβαλλοντική, αλλά συμβάλλουν και στη βιωσιμότητα των αλληλευτικών κοινοτήτων, γιατί χάρη στη συμμετοχή των γυναικών αυξάνεται το κατακεφαλήν ε, εισόδημα και χωρίς συμμετοχή των γυναικών θα ήταν κατάσταση πολύ πιο δεινή, ιδιαίτερα στα πλαίσια της κρίσης. Η συμβολή λοιπόν ε, της ε, αφανούς αυτής εργασίας των γυναικών σε ένα τόσο σκληρό τομέα όπως είναι η Ελία, η παρακλάδια του ελευτικού κλάδου, όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό το άδειλο λοιπόν αλλά ε, γενναίο έργο ήταν πολύ σημαντικό, γιατί οι γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες και αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες. Γιατί κάποιες ε, δουλειές, ε, όπως αυτές οι ιδιωτοκαλλιέργειες συγκέντρωσης μαλακίων και οστράκων, γίνονται αποκλειστικά και μόνο από τις γυναίκες, ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης. μερικές φορές είναι και κατά παράδοση γυναικείες τέτοιες δουλειές. Αλλά η κρίση απομάκρυνε τις γυναίκες και από αυτές τις θέσεις εργασίας, καθιστώντας ακόμη πιο επισφαλείς στις συνθήκες διαβίωσής τους. Διαπιστώνουμε λοιπόν από όλες τις μελέτες και τις εκθέσεις ε, που αναλύσαμε ότι υπάρχει ακόμη μεγάλη μισθολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. ιδιαίτερα εκεί που δεν υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις ε, όπως ε, στη μεταποιητική βιομηχανική οι γυναίκες λαμβάνουν 25% χαμηλότερους μισθούς από τους άνδρες. Και αποκλείονται πολλές φορές οι γυναίκες από τα διάφορα συστήματα διαχείρισης ε, των συνεταιρισμών, των μικρών επιχειρήσεων, των μικρών εταιριών και από τις επιχειρηματικές και εμπορικές οργανώσεις του ελευτικού κλάδου. Και παρά τις προσπάθειες που γίνονται εδώ και χρόνια ενισχύοντας ε, τα κυκλώματα των γυναικών προκειμένου να δημιουργηθεί μια αλληλεγγύη και άλλη υποστήριξη ε, θα πρέπει να έχουμε κατά νου αυτές τις ελλείψεις. Η πρώτη διάσκεψη που έγινε για το θέμα αυτό έλαβε χώρα το 2003, πριν από μια δεκαετία δηλαδή. Και η πρώτη πρωτοβουλία για την κατάσταση των γυναικών και ιδιαίτερα των κυκλωμάτων στήριξης των γυναικών έγινε το 2005 ήταν πρωτοβουλία μιας Βρετανίδας συναδέλφου, στην οποία θα ήθελα να αποτίσω φόρη τιμής, γιατί κατά κάποιο τρόπο κατάφερε να διαρρήξει ή να γεφυρώσει αυτό το κενό επικοινωνίας που υπήρχε στο Κοινοβούλιο. Έκτοτε σημειώθηκε σημαντική πρόοδος. Στη Γαλλικία ήρθα σε επαφή με γυναίκες που δουλεύουν στην υδατοκαλλιέργεια, στον πάλαμα των δεξιών, σε συνεταιρισμούς, ε, επιχειρηματίες, ασχολούνται με κοινοτικά προγράμματα, συμμετέχουν σε διάφορες ενώσεις και ισπανικές και πανευρωπαϊκές. Οπότε αυτή η όθηση που δόθηκε ήταν πολύ χρήσιμη και μάλιστα και κάποια κοινοτικά προγράμματα επέτρεψαν αυτή την οργάνωση των γυναικών σε δίκτυα και σε οργανώσεις και ήταν πολύ θετική η συμβολή τους. Είναι απαραίτητη και επίκαιρη και μια σχετική πρωτοβουλία τώρα για το θέμα αυτό και μάλιστα για την έκθεση στις παράκτες Ελίας, για την ΚΟΑ, για το Ταμείο. Ε, σήμερα το πρωί μιλήσαμε για την έκθεση του κ. Σαλαβράκου, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Συγκεντρώσαμε 31 τροπολογίες, αλλά την ώρα της αλήθειας και στις διαπραγματεύσεις, ε, στους τέσσερις τριμερείς διαλόγους, είχαμε μεγάλο πρόβλημα φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιοι ψυχολογικοί φραγμοί σε ό,τι αφορά την αναγνώριση μιας πραγματικότητας ε, και στα χαρτιά. Τελικά περιλήφθηκαν αρκετές τροπολογίες ε, για την ισότητα των φύλων και για την ε, μη διακριτική μεταχείριση, αλλά για να φτάσουμε στην θέσπιση κοινωνικών μέτρων και συγκεκριμένων ενισχύσεων, ώστε να ευνοήσουμε τις γυναίκες και μέσα από το, μέσα από το Ταμείο Αλίας και Θάλασσας, ή να χρηματοδοτήσουμε πολιτικές κατάρτισης για τις γυναίκες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ε, σε, στα ποικίλα καθήκοντα τέτοιων θέσεων επασχόλησης στην Αλία. Προσπαθήσαμε να τα προωθήσουμε όλα αυτά, εγώ από την ομάδα μου, τους σοσιαλιστές και δημοκράτες, αλλά σε τελική ανάλυση αρμόδια είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. θα είναι χρήσιμη η μελλοντική δημόσια ακρόαση με το θέμα αυτό για να ακούσουμε ένα φάσμα απόψεων και εμπειριών. Σημειώστε λοιπόν τη 14η Οκτωβρίου. Επίσης περιμένουμε και τη νέα μελέτη αξιολόγησης, ε, γιατί από το 2000 μέχρι σήμερα δεν είχαμε καμία ενημέρωση για το πώς, ε, την πρόοδος ε, συνέβη στο θέμα αυτό. Διάγνωση έχει γίνει, έχει μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα. Καλό θα ήταν και τώρα που έχουμε τους κανονισμούς και που διαρωτόμαστε τι μέλη να κάνουμε μια αποτίμηση της κατάστασης. Κατά τη γνώμη μου, όλες αυτές οι πτυχές που συγκεντρώνω αριστερά και δεξιά και ελπίζω να με βοηθήσετε κι εσείς ε, για να συμπεριλάβω στην έκθεσή μου, γιατί όλες οι καλές ιδέες χωράνε στην έκθεση αυτή, θα βελτιώσουν την συμμετοχή των γυναικών στον τομέα αυτό. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις εργασιακές τους συνθήκες, τα συμβόλαιά τους, τις αμοιβέ τους, να εξισωθούν με τις ε, αμοιβέ των ανδρών, να γεφυρωθούν οι μισθολογικές διαφορές, επίσης να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής και να ισχύσει ο κανόνας ίσα δικαιώματα για α, ίσες υποχρεώσεις, για αντίστοιχε υποχρεώσεις. Κατά τη γνώμη μου, η έκθεση αυτή δεν είναι μία τυχαία έκθεση πρωτοβουλίας. Είναι μία έκθεση πρωτοβουλίας που από την αρχή κρίναμε ότι είναι νευραλγική σημασία. Και ε, μερικές φορές όταν προσέκρουσα σε άγνοια ή έλλειψη κατανόησης προσπάθησα να την παραβλέψω. Περιμένω λοιπόν τα σχόλιά σας για να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα απαριθμεί με σαφήνεια τους στόχους, της καταθετήρες γραμμές, από όλα τα κοινοτικά όργανα και από τα κράτη-μέλη προκειμένου να αναγνωριστεί ο σημαντικό ρόλο των γυναικών σε ένα πολύ σημαντικό τομέα. Ναι και εγώ πολύ σύντομα γιατί είχαμε μιλήσει, έχω μιλήσει με την εισηγήτρια το θέμα αυτό το εκπονεί και η Επιτροπή Γυναικών επαναλαμβάνω ότι θέλουμε να συνεργαστούμε για την έκθεση αυτή Ξέρω τον ηγετικό ρόλο που έχει παίξει η, η συγγήτρια. Εμείς λοιπόν θα παίξουμε συντροματικό ρόλο για να ληφθεί υπόψη η οπτική γωνία της Επιτροπής Γυναικών και στο μέλλον θα έχουμε διάφορες ευκαιρίες για να το συζητήσουμε και φυσικά κατά την ακρόαση θα ε, εκφράσουμε την άποψή μας ε, για διάφορες παρεμβάσεις που θα Κυρία Μπιλμπάου, ευχαριστώ. Και εγώ στηρίζω την κυρία Ιέρο. Η ομάδα μας και εγώ θα παρακολουθήσουμε με θετική ε, και συνεπή στάση την προσπάθεια αυτή και γι' αυτό είχαμε υποβάλει και τροπολογίες στην ε, έκθεση Φερέρα για την ε, αλία βάθους Θέλουμε να μελετήσουμε τη συμβολή των γυναικών στον τομέα αυτό για την διατήρηση του τομέα, αλλά αυτό δεν έχει αναγνωριστεί. Γιατί ιδίω στην ε, μικρή κλίμακα αλληλεία οι γυναίκες συμμετέχουν στις οικογενειακέ επιχειρήσεις και η εργασία τους τουλάχιστον γινόταν για να μειωθεί το κόστος. Δηλαδή είχε οικονομική επίπτωση η εργασία τους. Και οι συστάσεις της μελέτης του 2008 που έλεγε ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε το ρόλο των γυναικών πρέπει να συνεχιστεί με τις χρηματοδοτήσεις των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων να επιμείνουμε στην κατάρτιση, ούτως ώστε στη συγκυρία τη κρίση, ή λόγω τη αναδιάρθρωση που βλέπουμε σε τόσους τομείς να μπορέσουν να βρουν άλλες δουλειέ, να αναγνωρίσουμε επαγγελματικά κάποιες δραστηριότητε του που αυτή τη στιγμή δεν αναγνωρίζονται σε διάφορα και να αναγνωρίσουμε τις ειδικέ ε, ε, νόσους αυτών των γυναικών ω επαγγελματικές νόσου. Όσοι ζούμε σε τέτοιο περιβάλλον ξέρουμε ότι οι γυναίκες των οικογενειών αυτών, οι γνωστές μας, ξέρουμε τι προβλήματα έχουν. Οπωσδήποτε, μετά από τόση προσπάθεια και τόσα χρόνια, δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί αυτές οι ασθένειες ότι σχετίζονται συγκεκριμένα με κάποια οικονομική δραστηριότητα. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε συνεπείς με τη στάση μας στο παρελθόν για τις διάφορες εκθέσεις και θα το κάνουμε, θα υποβάλουμε τροπολογίες για να αποδοθεί δικαιοσύνη στις ε, μητέρες και τις ε, γιαγιάδες μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, συζητήσαμε πριν από δύο χρόνια περίπου και στην Επιτροπή Γεωργίας κάτι πολύ παρόμοιο. Και διαρωτώ με, τι θέλετε κυρίες μου, πού στοχεύετε, τι θα ήταν τέλειο για σας. Και στην ουσία θέλω να θέσω τα εξής ερωτήματα. Πρώτον, αυτό που επιδιώκεται είναι απλώς να πείτε στις γυναίκες ε, στις χώρες σας ότι σας υποστηρίζουμε ή θέλουμε να υπάρξει νομοθεσία που θα πει στον τομέα πρέπει να απασχολήσετε περισσότερες γυναίκες. Τουλάχιστον οι Βρετανοί οι ψαράδες ε, δεν θα το έβλεπαν με πολύ θετικό μάτι. Πολλές φορές τα πληρώματά τους είναι οικογενειακή υπόθεση και παραδοσιακά ξέρω ότι μπορεί να με κατηγορήσετε ότι είμαι φαλοκράτης αλλά παραδοσιακά η γυναίκα μένει στο σπίτι και ασχολείται με τον οικοκυριό και οι άντρες ε, βγαίνουν στη θάλασσα και κινδυνεύουν. Θέλετε να τα αντιστρέψετε όλα αυτά. Θέλετε, τι, τι, ποιος είναι ο στόχος σας. Στόχος. Θέλετε νομοθεσία ή απλώς ε, να υποστηρίξετε. Και τι νομοθεσία. Θα χρησιμοποιήσετε λουκούμι ή βούρδουλα. Τι θα πείτε στους ε, καπετάνιους. Αν βάλετε περισσότερες γυναίκες στο πλήρωμά σας ε, θα πάρετε κάποια χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Ταμείο ή θα πείτε αν δεν βάλετε θα σας μειώσουμε την ποσόστοσή σας στη Γεωργία καταλήξαμε γιατί οι Γεωργοί πρέπει κάθε χρόνο να υποβάλουν ε, κάποια έντυπα. Πριν από δύο χρόνια ε, τα έντυπα αυτά ε, είχαν μια σειρά από ερωτήματα για το πόσες γυναίκες απασχολείται. Μήπως θα γίνει θέμα πολλαπλής συμμόρφωσης. τελικά βέβαια αυτό ξεθύμανε στον τομέα της Γεωργίας. Μήπως μπορείτε να μου πείτε σε 10 χρόνια πού νομίζετε ότι θα έπρεπε να έχουμε φτάσει με το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Όχι, όχι. Θέλει να πει τίποτα η Επιτροπή. Παρακαλώ. Είναι καθοδόν ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. Bueno, señor presidente. Ιέρο. Ε, πραγματικά ε, έμεινα άναυδη. Αυτή η απάντηση δεν δείχνει κανένα σεβασμό. Όχι, δεν επιδιώκω το τέλειο, αλλά σε κάποια σοβαρότητα και επίσης δεν είμαι ε, προφήτης, δεν ξέρω τι θα γίνει σε 10 χρόνια. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν οτροπίες σαν τη δική που αρνείται τα ίσα δικαιώματα και τις ίσες ευθύνες στις γυναίκες που έχουν και οι άνδρες σε όλους τους τομείς. Αυτό προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Θέλουμε να βελτιωθεί η κατάσταση όπου ενώ διαπιστώνουμε ότι είναι ενεργό και παραγωγικό τμήμα της δραστηριότητας η γυναίκα, δεν αναγνωρίζεται ο ρόλος της. Νομίζω να έχουμε καταλήξει σε 10 χρόνια σε ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες. Ευχαριστώ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα. Παρακαλώ. Ο κύριος Άγνιου, θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις παρούσες κυρίες ότι εγώ δεν πρόκειται να ε, υποβάλω υποψηφιότητα για, νερά, γοργόνα. Ε, μα δεν θα σας το και κανείς. Νομίζω ότι υπάρχει μια παροιμία στην Ισπανία που λέει ότι δεν ε, ε προσβάλλει αυτός που θέλει, αλλά αυτός που μπορεί. Ας το αφήσουμε εκεί. Επόμενο θέμα, 15. Απαγόρευση ε, εισαγωγών μεγαλόφθαλμου τόνου από ορισμένε χώρε. Είναι ο κανονισμό 1037 ε, του 2001. Υπάρχει μια πρόταση ε, κανονισμού, την πήραν οι πράσινοι και να δώσω το λόγο στον κύριο Ρωμέβα που είναι ο εισηγητής πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ακούσω την άποψη της Κομισιόν για να αντιδράσω. Καλύτερα να του ακούσω και μετά να απαντήσω. Βεβαίως έχετε δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Έκανα λάθος. Έχετε δίκιο. Η Βερόνικα Μπέιτς, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να μας παρουσιάσει την πρότασή της. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος. Καλησπέρα, Πρόεδρε. Καλησπέρα σα. Ε, είμαι πολύ ευχαριστημένη που για μια φορά η Κομισιόν μπορεί πρώτη να πάρει το λόγο. Ο τίτλο αυτού του σημείου είναι πολύ μακρύ, αλλά εγώ θα είμαι σύντομη και είμαι βεβαία πω αυτό το θέμα είναι λιγότερο επίμαχο από ό,τι το προηγούμενο. Τουλάχιστον ελπίζω να είναι. Η πρόταση αυτή είναι ε, καθαρά θέμα μεταγραφής μιας διεθνούς απόφασης που ελήφθη στην ICAT, ε, τη Διεθνή Επιτροπή για τη Διατήρηση των θερνοειδών του Ατλαντικού. «1827 ε, του 2008 ήταν η εφαρμοστική διάταξη για την εφαρμογή της απόφασης ICAT του 2004 για επιβολή απαγόρευσης εισαγωγών προϊόντων της ε, τον ε, τόνου που προερχόταν από την ε, ε, Βολιβία, Σιεραλεόνε κτλ. Αυτή η απόφαση, αυτός μάλλον ο κανονισμός εγκρίθηκε το 2005 ενώ η ΆΙΚΑΤ ήρε την απαγόρευση για την Καμπότζη, την ε, σημερινή Γουινέα και τη Σιέρα Λεώνα το 2005. Τώρα λοιπόν το 2011 η ΆΙΚΑΤ έλαβε άλλη υπόφαση και ήρε την απαγόρευση εισαγωγών για την Βολιβία και την... Ε, Ποια... τη Γεωργία. Λοιπόν, ε, πρόκειται απλά για μεταγραφή αυτή τη απόφαση, εφόσον έχει έρθει η απαγόρευση για όλε αυτέ τι χώρε και κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζεται να συζητηθεί περαιτέρω. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, Ωραία. Καλύτερα να δίνουν πάντα το λόγο στην Κομισιόν στην αρχή πάντα. Ε, ο Συμφωνώ με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα απλό κείμενο μετά της ε, εφαρμογής νομοθεσίας. Ε, θα συνεχίσουμε την ε, μέχρι τώρα παράδοση για τέτοιου είδους κείμενα και δεν ξέρω αν θα κάνουμε επευκαιρία και μια συζήτηση επί της ουσίας, αλλά ως προς το νομοθετικό πλαίσιο εμένουμε στην πολιτική που ακολουθούμε για τέτοιου είδου περιπτώσεις. Η κυρία Πατράου. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι όντω πέρα από ότι πρόκειται για μια απλή μεταγραφή μια συμφωνία, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να επιστήσουμε την προσοχή σε κάποιε πτυχέ που ξεχνάμε να τονίσουμε. Μία από αυτέ έχει να κάνει με το γεγονό ότι με αυτό το παράδειγμα βλέπουμε ότι αξίζει τον κόπο να επιβάλλονται κυρώσεις στις χώρες που δεν ε, πληρούν ε, τις ε, συμβάσεις και τις χώρες που ασκούν παράνομη και λαθρέα αλληλεία γιατί αποζημιωνόμαστε. Είναι δυνατόν δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει συμπεριφορές και με έναν διπλωματικό τρόπο να επιβάλλει τις καλές πρακτικές σε χώρες που αρχικά δεν τις ασκούσαν. Ήθελα αυτό λοιπόν να το τονίσω για την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε την έκθεση του κυρίου Ρωμέβα ακριβώς σε σχέση με την λαθρέα αλληλεία ε, και πάντοτε για αυτό το θέμα βλέπω πως ισχύει μεγάλη αυστηρότητα από πλευρά της Κομισιόν όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Στόλο, αλλά σπανίως ε, το ίδιο επίπεδο αυστηρότητα ισχύει για τρίτες χώρες και φαίνεται μάλιστα ότι κάποιες φορές η Κομισιόν φαίνεται σαν να είναι άοπλη, να μην έχει μέσα στη διάθεσή της για να επιβάλλει τους νόμους της σε τρίτες χώρες. Ενώ βλέπουμε πως στην ουσία έχει δυνατότητες που αν χρησιμοποιηθούν ε, ε, συνετά ασκούν επαρκή πίεση. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα. Ε, δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, επειδή μιλάμε για τον τόνο και για τρίτες χώρες, είναι και μιλάμε για την άρση της απαγόρευσης αγωγών, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως θα πρέπει να έχουμε μια γενική εικόνα του, τομέα, λευτικού τομέα της Ευρώπης και σε αυτή τη φάση όταν μιλάμε για αλίευση τόνου, για μεταποίηση, για βιομηχανία όλοι ανησυχούμε βεβαίως για τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Ταϊλάνδη και με τις δυνατότητες της ε, βιομηχανίας κονσερβοποίησης της Ταϊλάνδης που έχει να έρθει τώρα ε, να πλημμυρίσει τις αγορές μας με ε, πολύ φτηνά προϊόντα και έτσι να πνίξει τη δική μας βιομηχανία. Για να μην μου πείτε ότι είμαι εκτός θέματος, να μην ξεχνάμε ότι σε σχέση με την Ταϊλάνδη συχνά αυτό το ψάρι το οποίο ε, κυκλοφορεί σε κονσέρβες ε, πολλές φορές έχει αλλιευθεί χωρίς, καμία, χωρίς ε, ανευτήρησης καμιάς νομοθεσίας. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον τομέα και να μιλήσουμε, και εδώ μιλάμε για άρση της απαγόρευσης εισαγωγής τόνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχει άλλη παρέμβαση. Οπότε... Ολοκληρώνεται αυτό το σημείο και περνάμε στο επόμενο, το 16. Πρωτόκολλο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας Ακτής του Ελεφαντοστού. Α, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε που μου ξαναδίνετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα πολύ σύντομα να επανέλθω στα όσα είπε η βουλευτής για την παράνομη λαθρέα αλία. Να διευκρινίσω ότι αυτός ο κανονισμός δεν, ε, ε, ε, δεν απορρίπτει, δεν ακυρώνει τον κανονισμό IUU. Η Βολιβία και η ε, Καμπότζη έχουν συνυπογράψει αυτήν την νομοθεσία. Η άρση του εμπάργου από, υπό την ΆΕΚΑΤ δεν σημαίνει πως αυτές οι χώρες τώρα επιτρέπεται να εισάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μας ε, απαγόρευση εισαγωγών από την Γεωργία και την Πολυβία ε, υπό τον κανονισμό της Ένωσης παραμένει ανέπαφος. Αυτό για να διευκρινίσω το θέμα. Ευχαριστώ την Επιτροπή για το σχόλιο αλλά είναι άσχετο με αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν θέλει άλλο κανεί το λόγο, οπότε ολοκληρώνουμε το 15 και περνάμε στο 16. Πρωτόκολλο μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δημοκρατία τη Ακτή του Ελεφαντοστού σχετικά με το καθορισμό των αλληλευτικών δυνατοτήτων και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη Συμφωνία Αλληλευτική Σύμπραξη μεταξύ των δύο μερών. Ξέρετε, ω προ την εντολή του Συμβουλίου, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε διαπραγματεύσει με την ακτή του Ελεφαντοστού, προκειμένου να ανανεωθεί το πρωτόκολλο τη ε, Συμφωνία ε, σύμπρεξη και να παραταθεί για πέντε χρόνια από την 1η Ιουλίου του 2013. Την έκθεση ανέλαβε ο κύριος Κοτινή στον οποίο και θα δώσω το λόγο μετά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως που θα μας παρουσιάσει τις λεπτομέρειες της ε, συμφωνίας αυτής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με ιδιαίτερη χαρά θα σας ε, δώσω κάποιες διευκρινήσεις για αυτό το νέο πρωτόκολλο της Συμφωνίας Ελευτικής Σύμπραξης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ακτής του Ελεφαντοστού. Το νέο πρωτόκολλο μονογράφηκε τον ε, Ιανουάριο φέτος ε, και έχει πενταετή διάρκεια. Πρόκειται για μια συμφωνία που αφορά την αλίευση τόνου, σημαντική συμφωνία και στρατηγικής σημασίας για τον Ευρωπαϊκό Αλλιευτικό Στόλο, μια και είναι μεγάλη σημασία του λιμανιού της Αμπιτζάν για τη θυναλίευση, γιατί εκεί γίνονται εκφορτώσεις μεγάλων ποσοτήτων τόνου στη Δυτική Αφρική μέσω του λιμενιού της Αμπιτζάν. Ήταν σημαντική λοιπόν η ανανέωση της συμφωνίας και του σχετικού πρωτοκόλου με τη δημοκρατία της ακτής του Ελεφαντοστού. Ε, Επίση, ε, μην ξεχνάτε ότι το λιμάνι του Αμπιτζάν ζει από τις εκφορτώσεις τόνου και μάλιστα 20.000 άτομα ε, εκτιμάται ότι απασχολούνται ε, και εξαρτώνται άμεσα από την ε, Συμφωνία ε, Αλληλευτικής Σύμπραξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ακτή του Ελεφαντοστού. Ήταν απαραίτητη λοιπόν η ανανέωση της συμφωνίας και για την ακτή του Ελεφαντοστού για να εξασφαλιστούν οι εκφορτώσεις στο λιμάνι της Αμπιτζάν και όχι αλλού, αλλά είναι σημαντικό και για το δικό μας την αλληλευτικό τόνο, γιατί έτσι έχουμε ε, πρόσβαση και στις εγκαταστάσεις για εκφόρτωση του λιμανιού της Αμπιτζάν αλλά και στη μεταπι... στις μεταποιητικές μονάδες. Οπότε ε, ήταν επωφελής και για τις δύο πλευρές ε, η ανανέωση του πρωτοκόλου και της συμφωνίας. Ό,τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου πρωτοκόλου που μονογράφηκε τον Ιανουάριο, υπάρχουν αλληλευτικές δυνατότητες 28, για 28 τράτες και 10 παραγαδιάρικα. Έγινε μια μικρή τροποποίηση σε σχέση με τις ελευτικέ δυνατότητες που προέβλεπε το προηγούμενο πρωτόκολλο. Εκεί είχαμε 25 τράτες. Έχουμε μια μικρή αύξηση των τρατών ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τον αριθμό των τρατών που αλλιεύουν εκεί. Οπότε με τις 28 μηχανότρατες ευθυγραμμιζόμαστε με πολλά πρωτόκολλα με χώρες της περιοχής. Για τα παραγαδιάρικα είναι λίγη η παρουσία τους ε, και στο προηγούμενο πρωτόκολλο, γι' αυτό και τώρα μειώθηκαν ακόμη περισσότερο. Από 15 έχουμε 10 παραγαδιάρικα. Τώρα, ε, ως προς τα χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης κοινής ελευτικής πολιτικής ε, και αυτά αντικατοπτρίζονται στο νέο πρωτόκολλο, ρήτρες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές αρχές για παράδειγμα, αποσύνδεση ε, της πρόσβασης και της ατομιακής ε, συνδρομής και σημαντικό είναι να επισημάνουμε και την αύξηση της προκαταβολής που δίνουν οι εφοπλιστές. Και εκεί έλαβαμε υπόψη τις ε, συστάσεις και αποφάσεις της κοινής ελευτικής πολιτικής, της νέας κοινής ελευτικής πολιτικής την Καμπόν και τις αιχέλες, ίσως αλλάξει το μοντέλο, αλλά ήδη διαπιστώνουμε μια αύξηση κατά 40% των προκαταβολών που καταβάλουν οι εφοπλιστές. Σε ό,τι αφορά τα αλλιευτικά αποθέματα, είναι τα τρία είδη τροπικού τόνου που αλλιεύονται. Αλβακόρ, Λιστάο και Πατό είναι ελευτικά αποθέματα σε καλή κατάσταση. Η αξιολόγηση γίνεται από το ICAT, τη Διεθνή Επιτροπή διατήρηση των θηναλευτικών αποθεμάτων και ε, ακολουθούμε φυσικά και τις συστάσεις του ΙΚΑΤΣ ότι αφορά τον προσδιορισμό των ε, ποσοστός, των ποσοτήτων. Τώρα, η χωρητικότητα αναφορά πέρασε από 7.000 σε 6.500 τόνους, λαμβάνοντας υπόψη και τη προηγούμενη συμφωνία και κρατώντας ένα αρκετά υψηλό επίπεδο χωρητικότητας, ε, δεδομένης της ιδιαιτερότητας αυτής της χώρας. Το 2010-2011 η χώρα πέρασε από μια δινή κρίση, έμοιαζε σχεδόν με εμφύλιο πόλεμο, οπότε τότε οι ελευτικές μας δραστηριότητες μειώθηκαν, ουδέποτε δεν σταμάτησαν, αλλά μειώθηκαν δραστικά, επηρεάστηκαν από την πολιτική κατάσταση στην ακτή του ελεφαντοστού. Οπότε προβλέψαμε ένα περιθώριο μεταξύ των ε, ε, τωρινών και των μελλοντικών αλληλευτικών προσπαθειών που θα αυξηθούν δεδομένου του, κρίσιμου, του κέριου ρόλου που διαδραματίζει το λιμάνι της Αμπιτζάν. Και τέλος, προϋπολογισμός 680 εκατομμύρια ευρώ. Μικρή αύξηση σε σχέση συγγνώμη, ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο πρωτόκολλο. 680.000 ε, ευρώ, ε, μια μικρή μείωση της πρόσβασης, ε, μια και μειώθηκε και η χωρητικότητα αναφοράς, ενώ αυξήθηκε αισθητά η τομεακή συνδρομή. Εκεί περάσαμε από 140.000 σε 250.500 για την τομεακή συνδρομή λαμβάνοντας υπόψη τις μεγάλες ανάγκες ε, της χώρας αυτής ε, για ενίσχυση των μέσων ελέγχου και επιτήρησης. Γιατί η χώρα πέρασε από τεράστια κρίση, πρέπει να γίνει κάποια ανασυγκρότηση. Ε, οι αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση, δορυφορική παρακολούθηση των σκαφών, για τον έλεγχο και ούτω καθεξής. Βέβαια το χρήμα δεν είναι το παν και αποφασίσαμε να στηρίξουμε και με προσπάθεια δημιουργίας υποδομών ε, και με τεχνογνωσία τη χώρα αυτή και στείλαμε οι υπαλλήλους μας στην Αμπιτζάν για να προσφέρουν ε, έμπειρο γνωμοσύνη και τεχνογνωσία στις ε, αρμόδιες αρχές της ακτής του Ελεφαντοστού για να καταπολεμήσουν την παράνομη λαθρέα και άναρχη και να βελτιώσουν τη διαχείριση των αλλιευτικών τους πόρων. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσης. Επίση, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Δημοκρατία του Ελεφαντοστού, που είναι ένας εταίρο πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα στην ε, περίοδο της κρίσης ε, εμείς ε, αδιάλειπτα στηρίξαμε την κυβέρνηση, στηρίζαμε την κυβέρνηση του κ. Γουαταρά. Οπότε η συμφωνία αυτή ευθυγραμμίζεται με τη γενική μας πολιτική προσέγγιση απέναντι στη δημοκρατία της, της ακτής του Ελεφαντοστού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κ. Σκοτεινή.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 Επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να αναφέρω κάποιες σκέψεις στο πρωτόκολλο που ορίζει τις δυνατότητες ε, της αλληλευτικής και τη συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την ακτή του Ελεφαντοστού. Ε, εκπνέει το καλοκαίρι και η νέα συμφωνία προβλέπεται για πέντε έτη και ισχύει από την εκπνοή του ισχύοντος ε, πρωτοκόλλου. Μετά από, μάλλον τρέχοντας, θα έλεγα ότι αυτή η συμφωνία είναι ισορροπημένη. Γενικά εξασφαλίζεται μια επαρκή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανάπτυξη αλίας στην ακτή του Λεφαντοστού, στη μεταβατική περίοδο που διανύει αυτή τη στιγμή η χώρα, καθώς ε, και μια αποδοτική ε, λύση για, την ευρωπαϊκή, για τον ευρωπαϊκό στόλο. Είναι μια συνενετική συμφωνία που ε, βρήκε ε, που είχε αίσια έκβαση μετά από δύο γύρους μόλις διαπραγματεύσεων, πράγμα που οδηγεί στο ότι να εννοήσουμε ότι οι δύο πλευρές είναι ευχαριστημένες. Είναι μια συμφωνία που δείχνει την καλή διακυβέρνηση της Ένωσης. Ε, βέβαια, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορεί να αποτελέσει περίπτωση όπου θα ανασταλεί η ισχύ της ε, συμφωνίας. Περιλαμβάνονται οι σχετικές διατάξεις όπως στις περισσότερες διμερείς αλληλευτικές συμφωνίες στην περιοχή. Υπάρχουν προβλήματα προβλέψεις ε, για επιχειρησιακή ε, χρήση του ηλεκτρονικού ημερολογίου πλοίου για το 2014. Από την άλλη πλευρά, από πολιτική άποψη, είναι μια συμφωνία που πρέπει να δείξει τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και κυρίω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μια χώρα που βγαίνει από τον εμφύλιο και που ε, μπαίνει στην πορεία τη δημοκρατία και τη συμφιλίωση. Η εκτή του λεφαντοστού είναι υπό ανοικοδόμηση, υπό ανασυγκρότηση και πρέπει να ολοκληρωθούν διάφορα έργα. Το μεγάλο εργοτάξιο του πολιτικού διαλόγου προχωρά. Ε, έχει ξεκινήσει πολιτικό διάλογο με την αντιπολίτευση, δημιουργία μια εναρμόνιση διαλόγου, αλήθεια συμφιλίωσης, ε, του οποίου προεδρεύει ο Σάλκον Μπανί και προχωρά προς την κατεύθυνση. Έχουν επίσης γίνει πρόοδοι ε, με την πρόσφατη απελευθέρωση Λουρά Ακούν που είναι ο ε, γραμματέας του Λαϊκού Μετόπου της Ακτής του Ελεφαντοστού. Δείχνουμε τη στήριξή μας και στον Πρόεδρο Βάταρα, ε, μια στήριξη σε αυτή τη χώρα που είναι υποπλήρη ανασυγκρότηση και νομίζω πως αυτή η συμφωνία θα πρέπει να έχει θετική ε, αντιμετώπιση από την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Κοτινή. Ο κύριος Βαουένσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω μια ερώτηση για το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου για τις ε, νέες ελευτικές άδειες ε, και τις ε, δηλώσεις στα πιστοποιητικά. Φυσικά γνωρίζουμε ότι αντικείμενο είναι ο τόνος και το, στο άρθρο 6 αναφέρεται ότι αν ευρωπαϊκά ελευτικά σκάφη ενδιαφέρονται για άλλες αλληλευτικές δραστηριότητες που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα έχει διαβουλεύσεις με τις αρχές της ακτής του Ελεφαντοστού για την πιθανή χορήγηση αδειών για νέες αλληλευτικές δραστηριότητες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω για τα πελαγικά, μικρά πελαγικά είδη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον που υπάρχει και για αυτού του είδους στην Αλία. Gracias, Uh, thank you very much uh, for the presentation. Ευχαριστώ για την παρουσίαση. Πολύ θετικό ότι οι αρχή της νέας ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής εφαρμόζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ε, αποσύνδεση κτλ. Μία ερώτηση. Οι καρχαρίες ως παραλίευμα. Το πρωτόκολλο με την ε, Μαδαγασκάρη υπήρχε ένα πολύ θετικό στοιχείο. Πρώτη φορά σε ένα τέτοιο πρωτόκολλο αναφέρονταν εκπεφρασμένα οι καρχαρίες. Και αν δούμε τα αλλιεύματα, οι καρχαρίες είναι 50 και πάνω της 100 των αλλιευμάτων. Υπάρχουν προβλέψεις ε, για τους καρχαρίες σε αυτό το πρωτόκολλο. Και αν όχι, γιατί όχι. Και αύξηση της αμοιβή των πλειοκτητών. Των τελών για τους πλειοκτήτες. Γιατί αυξήθηκαν. Να μας εξηγήσετε παρακαλώ λίγο καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρος. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για αυτές τις ερωτήσεις. Για το θέμα των άλλων ειδών. Υπάρχει μηχανισμός για να αλλιευθούν. Αλλά θα έπρεπε να τηρούνται μια σειρά προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα διαβούλευση με τη χώρα και δεύτερον η κατάσταση των αποθεμάτων να επιτρέπει τη δυνατότητα αλήψης των πελαγικών ή άλλων ειδών. Και τρίτη προϋπόθεση, να τροποποιηθεί ε, προς αυτή την κατεύθυνση το πρωτόκολλο. Γιατί στο άρθρο 1 αναφέρονται τα ε, ιδιαίτερα αποδημητικά είδη προβλέπονται οι δυνατότητες αλλά με βάση κάποιες προϋποθέσεις και φάσεις που πρέπει να διανυθούν πριν ανοίξει το πρωτόκολλο και σε άλλα είδη. Για τους καρχαρίες. Ο ευρωπαϊκός στόλος ε, στις ακτές ε, της ακτής ελεφαντοστού δεν επιδιώκει να αλλιεύσει αυτά τα ψάρια. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από τη Μαδαγασκάρη. Τα παραγαδιάρικα δεν είναι κατάλληλα για να ψαρέψουν στην ε, ε, οικονομική ζώνη της ακτής ελεφαντοστού και γενικότερα στη Δυτική Αφρική. Είναι διαφορετική κατάσταση λοιπόν εδώ σε σχέση με άλλες συμφωνίες. Για την ε, οικονομική λογική δεν θίξαμε την τιμή αναφορά στον 100 ευρώ τον τόνο, 35 πληρώνουν οι πλειοκτήτες και 65 η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει μια διαφορά ε, για τις προκαταβολές. Οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές που θέλουν, που θέλουν να αλλιεύσουν στην ε, ακτή λεφαντοστού πληρώνουν περισσότερα, πάνω από 40%. Εδώ για παράδειγμα για τις στράτες 5.000 και άλλο ποσό για τα παραγαδιάρικα. Αυτό είναι μια εγγύηση εισοδήματος και παρουσίας ε, ε, στα ύδατα της ακτής Λεφαντοστού. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία, λέει ο πρόεδρος. Άλλες παρεμβάσεις? Όχι. Ωραία. Έληξε εσείς για το θέμα αυτό. Το επόμενο... Ε, ε, θέλει κανείς να πει τίποτα. Τώρα, για τη συμφωνία των συντονιστών έγινε η κατανόμη των εκθέσεων, των γνωμοδοτήσεων. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, εγκρίνουμε τις αποφάσεις των συντονιστών και περνάμε στο τελευταίο σημείο, επόμενη συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου, όπως ξέρετε, πρωί και απόγευμα και 11 Ιουλίου το πρωί μόνο. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς το λόγο. Κύριος Άγνιου. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Σημείο 17. Τι έπαθε, τι συνέβη, δεν το συζητήσαμε. Τι έγινε, αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Ναι. Όταν εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη, χθες, σας ενημέρωσα ότι και το σημείο 14 και το σημείο 17 αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση του Ιουλίου. Έτσι εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη με δύο αναβολές περνάει το 17 στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Οπότε αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, λύεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ θερμά όλους και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Ναι,